Buenas tardes a todos. Creo que... Καλησπέρα σα, λέει η πρόεδρο. Les doy la bienvenida a la reunión del Comité LIBE en videoconferencia. Les agradezco... Δεν ακούω. καλωσορίζουμε λοιπόν σε αυτή την τηλεδιάσκεψη και θα σα ευχαριστήσω εκ βάθου καρδιά formación técnica. También les ruego, durante el tiempo de la sesión, que... Αυτός είναι ο χρόνο που έχουμε και πρέπει όπως και τις άλλες φορές να δείξουμε υπομονή. Γιατί τα εργαλεία που έχουμε να δουλέψουμε δεν είναι και τέλεια. Οπότε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, πέστε το και κάποιο τεχνικό θα σα βοηθήσει. Θα πρέπει επίση να σα πω ότι θα πρέπει να κάνουμε δύο συναντήσει των δύο ώρων, γιατί έτσι θα μπορέσουμε να μειώσουμε τον κίνδυνο για αυτού που βρίσκονται στο Κοινοβούλιο, ούτω ώστε να εξασφαλίσουν την διεξαγωγή τη συνάντησή μα. Και αυτό αφορά και την ομιλούσα. Επίση, θα πρέπει να σα πω ότι από πλευρά διερμηνία έχουμε έξι γλώσσε. Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά, ελληνικά και γερμανικά. Μας αναφέρουν οι διερμηνείς ότι η ποιότητα εικόνας και ήχου είναι σημαντική, ούτω ώστε να μπορέσουν να εξασφαλίσουν το ότι θα περάσει το μήνυμα. Και σας ε, παρακαλούν να ακολουθήσετε τους κανόνες που προβλέπονται για την σύνδεσή σας. Και θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι η τηλεφωνική σύνδεση δεν επιδέχεται διερμηνία. Επίσης και δεδομένων αυτών των συνθήκων παρακαλούμε όποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει την μητρική του γλώσσα και αυτό να το κάνει με έναν ρυθμό φυσιολογικό. Να μην διαβάζει γρήγορα χρησιμοποιώντας κάποιες σημειώσεις όπως συνήθως. Ιδίως δε να ευχαριστήσουμε τους διερμηνείς και όλους τους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Διερμηνίας. Και πάλι σας ευχαριστούμε που μας βοηθάτε να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη Ο πρόεδρος Χουάν Φερνάντο Λόπες Αγγιλάρ θα λάβει τον λόγο τώρα, ελπίζω να μπορεί. Μας ακούτε πρόεδρε, μας ακούτε, έχετε σύνδεση. Έχετε το λόγο. Και πάλι Μάιτε, γεια σου και σας ευχαριστώ που ήρθατε. Σας ευχαριστώ κυρία Αντιπρόεδρε για όσα έχετε κάνει. Οπότε ας ε, ξεκινήσουμε τώρα. Έχετε κάποια ένσταση για την διάταξη, όχι, επομένω εγκρίνεται. Και τώρα έχουμε το θέματα που πρέπει να ανακοινώσω. Δηλαδή θα πρέπει να εγκρίνουμε τα όσα προτείνουν οι ε, συντονιστές. Πάντως το θέμα αυτό αναβάλλεται για τις 12 Μαΐου και άρα τώρα θα πρέπει να σας πω ότι σήμερα θα πρέπει να κάνουμε ψηφοφορία. Η ψηφοφορία που θα γίνει με ψηφοδέλτια. Και από απόσταση δεδομένη της καταστάσεως. Οπότε αυτοί οι συνάδελφοι έχουν ε, λάβει ένα email που αναφέρει ότι ξεκινά η ψηφοφορία για τις ε, τροπολογίες του θέματος και πρώτα-πρώτα να δούμε αν έχουμε απαρτία. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ζητήσουμε από αυτούς που ζητούν τον λόγο να πατήσουν ένα κουμπί για να επιβεβαιώσουν την παρουσία τους ε, και αυτό έχει σχέση βέβαια με το software ε, αυτής της ιντερνετικής μετάδοσης. Επίσης, αυτοί που λαμβάνουν μέρος στην ψηφοφορία παρακαλούμε ή να τυπώσουν το ψηφοδέλτιο επί τη βάση της λίστας ψηφοφορίας και εκεί να συμπληρώσουν όνομα, ψήφο ή θα πρέπει να φωτογραφίσουν ή να σκανάρουν ε, εκεί που πρέπει με email ε, το ψηφοδέλτιο. Και όλα αυτά ως λίστες που θα σταλούν από την επίσημη διεύθυνσή σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Θα πρέπει όλα αυτά να είναι βανάγνωστα, να έχουν την υπογραφή σας και σας ε, υπενθυμίζω ότι έτσι θα έχουμε έγκυρη ψήφο και μόνο όσες ψήφοι ληφθούν σε αυτό το κουτί του ταχυδρομείου θα μετρήσουν, θα δώσουν έγκυρες. Οπότε μισή ώρα από τώρα θα έχει κλείσει η ψηφοφορία. Οπότε μόνο όσοι προλάβουν αυτή την προθεσμία θα ληφθούν υπόψη. Επίσης σας ενημερώνω ότι η πρώτη τροπολογία από τον συνάδελφο Ισαβέλ Λίμα και η δεύτερη τροπολογία του Νικόλα Προκατσίνη είναι ταυτόσιμες και άρα θα τις ψηφίσουμε από κοινού. Ε, στις 4 και 4 θα ανακοινώσουμε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αυτών των δύο τροπολογιών. Στη συνέχεια όμως, αφού τις ψηφίσουμε αυτές τις δύο που θα τις ψηφίσουμε από κοινού, ε, τότε θα ξανά ψηφίσουμε θα πρόκειται για την ψηφοφορία ε, του σχεδίου της γνωμοδοτήσεως και τελικά θα γίνει τελική ψηφοφορία στις 5 και μισή. 5.30 με 6.30 δηλαδή θα κρατήσει εκείνη η ψηφοφορία με την ίδια διαδικασία ψηφίσεως. Οπότε το αποτέλεσμα αυτής της τελικής ψηφοφορίας πρόκειται να κοινοποιηθεί στους συναδέλφους στις 8 και 55 δηλαδή 5 λεπτά ε, πριν κλείσει η απογευματινή μας συνεδρίαση. Θα ανακοινωθεί με email το αποτέλεσμα και θα καταχωρηθεί στα πρακτικά μας. Άρα, 5.30 με 6.30 η τελική ψηφοφορία και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μία ώρα αργότερα. Όπως ξέρετε είμαι ο εισηγητής, οπότε έχουμε τώρα να ψηφίσουμε την εκτελεστική απόφαση για έναξη αυτοματοποιημένης αλλαγής δακτυλοσκοπικών δεδομένων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό είναι το θέμα της ψηφοφορίας, η γνωμοδότηση. Και τώρα, σας προτείνω να προχωρήσουμε ε, στα θέματα ιστορικών υποθέσεων με το πρώτο ουσιαστικό θέμα για σήμερα. Ιστορικέ υποθέσει στην εποχή του COVID-19, θέματα χώρου έγκυνα σύλλου, μετανάστευση και ασφάλεια. Προβλέπεται ανταλλαγή απόψεων με την αρμόδια επίτροπο την Ήλβα Γιώχανσον. Χαίρομαι αγαπητοί επίτροπε που θα τα συζητήσουμε ακόμα και από αυτές τις συνθήκες και μέχρι ότου ξεπεράσουμε αυτή την κρίση του κορονοϊού θα πρέπει να διατυπώσουμε τις επιφυλάξεις μας σε σχέση με όλα αυτά τα θέματα που μας προβληματίζουν, μας ανησυχούν και όσον αφορά τα δικαιώματα που καλύπτει το θέμα μας. Και ενδιαφέρει πάρα πολύ την Επιτροπή να ζητηθεί η υπόθεση αυτή όσον αφορά την αναστολή του Σέγγεν Συγγνώμη, συγγνώμη πρόεδρε, λέει πρόεδρος, υπάρχει ένα θέμα τεχνικό. Παρακαλώ να ζητηθεί η επαλήθευση της ε, απαρτίας, γιατί μου λέει η γραμματεία ότι πρέπει να γίνει αυτό, να επαληθεύσετε αυτό με το αντίστοιχο κουμπί της ε, συμμετοχής της Ιντερνετικής. Χωάν Μάλιστα, εντάξει, το κατάλαβα, το κατάλαβα, λέει ο κύριος Λόπες Αγγιλάρ. Μάλιστα, μάλιστα. Εάν όλοι είναι σε θέση να το κάνουν, βλέπουν το κουμπί, έχουν το software, θα πρέπει εκεί να καταλάβουν ότι πρέπει να δηλώσουν ότι συμμετέχουν στη συζήτηση και άρα πρέπει να κάνουμε αυτήν την επαλήθευση της απαρτίας. Να το δούμε τώρα. Πρόεδρε, πρόεδρε, συγγνώμη, λέει η πρόεδρος. Ναι, ναι, έχουμε απαρτία, μπορείτε να συνεχίσετε. Α, μάλιστα, τότε έχουμε απαρτία. Και όπως είπα, τότε θα προχωρήσουμε στο θέμα ουσίας σημερινής συνεδρίασης. Αυτό θα πρέπει όμως να συζητηθεί με την Επίτροπο Ιωάννησον. Όπως είπαμε, είναι πάρα πολύ σημαντική η υπόθεση του Σένιερ που έχει ανασταλεί. Επομένως, δεν έχουμε ελεύθερη διακίνηση των προσώπων, κάτι το οποίο είναι ένας θησαυρό για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα σημαντικό εκτιμένο, αλλά είναι και τα θέματα του ασύλου, διότι είπαμε ότι έτσι θίξαμε το ζήτημα των στρατοπέδων, των καταβλισμών των μεταναστών, αλλά αυτό δεν είναι το μόνο θέμα. Επίσης, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει στην ε, Μεσόγειο, τι γίνεται με όλους αυτούς που θέλουν να μπουν από τα εξωτερικά σύνορα και τα οποία πιέζουν. Κάποια σημεία των εξωτερικών σύνορων τα πιέζουν. Συγκεκριμένα πιέζεται η Μάλτα, η Ιταλία, η Ισπανία, τα Κανάρια νησιά. Ο, και έχουμε περιοριστικά μέτρα αυστηρά στα Κανάρια νησιά και εκεί ε, υπάρχει απαγόρευση, υπάρχει αναστολή της ε, συνήθους διαδικασίας σε Κανάρια, σε νησιά. Παρ' όλα αυτά και στην Ισπανία, αλλά και έχουμε και το θέμα της Δυτικής Αφρικής, γιατί από εκεί ξεκινά ο κόσμος και πηγαίνει ε, στις ε, ακτές των ε, Καναριών νησιών υπό και επίσης θα πρέπει να συζητήσουμε τα θέματα ασφάλειας. Επομένως, έχουμε όλα αυτά και σας προτείνω να ακούσουμε τι έχει να μας πει επί ένα τέταρτο η Επίτροπος και να γίνει ένας πρώτος γύρος ερωτήσεων από τους ε, συντονιστές. Τρία λεπτά μάξιμο καθένας, οπότε να υπάρχει χρόνος για τους υπόλοιπους να λάβουν το λόγο και να πούν ό,τι θέλουν να πούν και να τους πει η Επίτροπος. Οπότε, ας αρχίσουμε. Αν μας ακούτε, Επίτροπε, έχετε το λόγο. So, hello everybody. Γεια σας με ακούτε, με βλέπετε. Καλησπέρα προς την Επιτροπή Λίμπε και χαίρομαι ιδιαίτερως που βρίσκομαι και πάλι μαζί σας. Θα αναφερθώ σε διάφορα ζητήματα και σε, διάφορα, σε πτυχές της κατάστασης της κρίσης του COVID. Όλοι περνούμε δύσκολους καιρούς. Η οικονομία, η απασχόληση, η υγειονομική περίθαλψη, είναι υπό μεγάλη πίεση και οι προβλέψεις είναι ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα περάσουμε στη πιο βαθιά κρίση και ύφεση που έχουμε περάσει ποτέ. Είναι τεράστια λοιπόν η πρόκληση αυτή. Πρόκληση σε ό,τι αφορά τα σύνορα, την ελευθερία μετακίνησης, όπως μόλις ανέφερε ο Πρόεδρος, αλλά οι προκλήσεις αυτές αφορούν και το θέμα του ασύλου και της ασφάλειας. Να ξεκινήσω με το σκέλος της ασφάλειας. Το οργανωμένο έγκλημα γρήγορα προσαρμόστηκε στην κρίση και οι εγκληματίες θα ε, χρησιμοποιήσουν και θα εκμεταλλευτούν την οικονομική ύφεση. Και έτσι λοιπόν το κυβέρνο έγκλημα μέσω της σεξουαλικής εκμετάλλευση των παιδιών και το κυβέρνο έγκλημα λοιπόν ε, δημιουργήθηκε προβλήματα στην Τσεχία σε ό,τι αφορά το ίντερνετ η ζήτηση για την σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών έχει αυξηθεί κατά 30% σε κάποια κράτη-μέλη, Πρόεδρε, και οι ευρωπαϊκές αστυνομικές δυνάμεις καταπολεμούν τους εγκληματίες μαζί με τις αρχές της Γερμανίας, της Ιρλανδίας, των κατοχωρών. Προσπαθήσαν λοιπόν να καταπολεμήσουν περιπτώσει απάτη ύψου 15 εκατομμυρίων με πλαστέ και ε, ανύπαρκτε ε, μάσκε προστασία. Ε, δεν μπορούμε να πούμε κάτι οριστικό για τα νέα αυτά μοντέλα που δημιουργούνται, αλλά πρέπει να καταπολεμήσουμε αυτή την ε, αυτό το έγκλημα, την καταπολέμηση, να καταλαβαίνουμε επίση τη σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών. Θέλουμε να υποστηρίξουμε τα θύματα και να αποφύγουμε την απομόνωσή του. Θέλουμε να ενισχύσουμε την εντολή τη Ευρώπη, να βελτιώσουμε την ανταλλαγή πληροφοριών για του εγκληματίε ό,τι αφορά το DNA, τα δακτυλικά αποτυπώματα. Θέλουμε να βοηθήσουμε τι αρχέ επιβολή του νόμου μέσω εκπαίδευση, μέσω τη τεχνολογία και σήμερα η Επιτροπή υποβάλλει ένα σχέδιο δράση για να καταπολεμήσει την χρηματοδότηση εγκληματικών δικτύων και την, ε, το ξέπλυμα χρήματο. Δεν είναι δυνατόν 1% του ΑΕΠ, πάνω από 100 εκατομμύρια, δισεκατομμύρια ευρώ από το οργανωμένο έγκλημα θα κατάσχονται. Θα πρέπει να δούμε να περιληφθούν μάλλον και τα έσοδα από το τράφικινγκ ανθρώπων. Δεν πρέπει να μειώσουμε την ε, καταπολέμηση των εγκληματικών αυτών δικτύων. Θα πρέπει να ε, δούμε και ποιες είναι οι νέες προκλήσεις. Ελπίζουμε αυτά, αυτές οι συμμορίες να μην χρησιμοποιήσουν και τον ιό και τα βιολογικά όπλα, σε ό,τι αφορά το σκέλος του ασύλου και τη μετανάστευση. Όλοι αντιμετωπίζουμε προκλήσει ασφαλώ. Το συζητήσαμε και την προηγούμενη φορά που συναντηθήκαμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει κατευθυντήριες γραμμέ για το πώ θα πρέπει να εκτελεχθούν διαδικασίε μετανάστευση και μετεγκατάσταση. Είτε έχουμε COVID είτε όχι, όλοι έχουν δικαίωμα ε, να έχουν πλήρη πρόσβαση στα δικαιώματά τους. Από την τελευταία φορά που μιλήσαμε, 12 ασυνοδευτοί ανήλικοι από τα στρατόπεδα της Ελλάδας έχουν πάει στο Λουξεμβούργο, 47 ε, στη Γερμανία. Και τώρα ετοιμαζόμαστε για τα επόμενα βήματα με τη Σλομανία και την Πορτογαλία. Θα συνεχίσουμε λοιπόν την μετεκατάσταση και θα είναι συνολικά 1.600 ασυνοδευτοί ανήλικοι που θα μετεκατασταθούν σε 10 κράτη-μέλη τους επόμενους μήνες. Επίσης προχωρήσαμε σε ό,τι αφορά την μετεγκατάσταση των πιο ευάλωτων ε, ομάδων από τις καταβλισμούς στα νησιά. Έχει ήδη ξεκινήσει η αντιδικασία αυτή και μίλησα με τον Έλληνα Υπουργό πριν από κάποιες ημέρες. Τα ευαίσθητα αυτά άτομα μεταφέρθηκαν εκτός των καταβλισμών ε, την ε, προηγούμενη εβδομάδα. Θα ακολουθήσουν 390 αυτή την εβδομάδα και την επόμενη εβδομάδα 600 τέτοια άτομα ευάλωτα. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι πολλοί καταφθάνουν πλέον σε βάρκες στη Μάλτα και στην Ιταλία. Ανησυχούμε για την ασφάλειά τους και πάλι η Ιταλία και η Μάλτα είναι αυτοί που ε, δέχονται πιέσεις. Στο πρώτο Συμβούλιο Ιστορικών Υποθέσεων στο ε, προηγούμενο μάλλον Συμβούλιο Ιστορικών Υποθέσεων, κάλεσα τα κράτη-μέλη να δείξουν αλληλεγγύη. Και βλέπουμε τεράστιες ε, πιέσει και στι Καναρίε νήσους. Τεράστιες πιέσει επίσης, λοιπόν, και εκεί στην παρούσα φάση. Όπως σα ανακοίνωσα και στην τελευταία συνεδρίαση τη Επιτροπή ΛΥΜΠΕ πριν από δύο ημέρε, ξεκίνησα μία συνάντηση με του. Ε, ε, Κοινωνικού εταίρου και τις οργανώσεις τη κοινωνία των πολιτών για να ακούσω τι λένε αυτοί για την υποστήριξη και την προστασία των μεταναστών στην κρίση αυτή του κορονοϊού και πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να αυξήσουμε την ε, οικονομική συμβολή στη φάση της ανάκαμψης. Ήταν πολύ καλή αυτή η συνάντηση και τις επόμενες εβδομάδες θέλουμε να κλείσουμε μια καινούρια ε, συνεργασία και τρική σχέση για την ανάκαμψη μετά την κρίση αυτή. Τρίτο θέμα, τα σύνορα. Μετά από την ε, κρίση, μετά το ξέσπασμα της κρίσης, πολλά κράτη-μέλη επανεσύγαγαν ελέγχους ε, στα σύνορα. Το θέμα αυτό δεν είναι τα σύνορα, λοιπόν. Είναι ο ιό. Γιατί και μέσα στα κράτη-μέλη, σε πολλέ περιπτώσει, ρισκάρει κανεί μεγάλο πρόστιμο αν επισκεφθεί φίλου ή αν φύγει το Σαββατοκυριακό. Και δέχομαι δεκάδε επιστολέ από απελπισμένου πολίτε και εσείς φαντάζομαι ως βουλευτές δέχεστε πολλές αρχές επιστολές με ερωτήσεις, με εκκλήσεις για βοήθεια. Οι πολίτες λένε είμαι στην Αυστρία, είμαι στην Ελλάδα, είμαι στην Πολωνία. Πώς θα επιστρέψω στη χώρα μου, στη Γερμανία, στη Βουλγαρία, στην Σλοβενία. Είμαστε συνταξιούχοι. Έχουμε κολλήσει σε μια άλλη χώρα. Πώς θα γυρίσουμε. Και στο Βέλγιο λέει για παράδειγμα κάποιος ότι έχω τον αραβωνιαστικό μου στην Γαλλία. Δεν μπορεί ο σύντροφό μου να έρθει να δει την κόρη του που μόλι γεννήθηκε. Πραγματικά σπάραξε κάρτε ιστορίε. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκδώσει ε, γραμμέ για να υπάρξει ροή ιατροφαρμακευτικών προϊόντων και να βοηθήσει τον κόσμο που εργάζεται σε άλλο κράτο μέλο. Να μειωθούν επίση ε, ε, ο ε, στα σύνορα. Στα σύνορα. Ε, κάναμε 12 τηλεδιασκέδεις με την ε, ομάδα του COVID, 6 υπουργικές συναντήσεις και πολλές διμερείς συναντήσεις. Η κατάσταση είναι πλέον ε, σταθερή. Δεν είναι όμως απαραίτητα ούτε βιώσιμη για το μέλλον, ούτε αποδεκτή. Προφανώ ο κόσμος είναι εξοργισμένος, απελπισμένος, αγανακτισμένο, γιατί έχουμε διαπιστώσει έτσι πόσο έχει γίνει αναπόσπαστο τμήμα τη ζωή μα η ελεύθερη μετακίνηση. Κάποιε φορέ χρειάζεται να μα πάρουν κάτι για να καταλάβουμε πόσο το εκτιμούμε. Και έτσι ο COVID μα δείχνει πώ θα ήταν η Ευρώπη χωρί ελεύθερη μετακίνηση. Πολλά εκατομμύρια αμα, πολίτες στην Ανατολική και την Κεντρική Ευρώπη θυμούνται πώς ήταν να είναι αποκλεισμένος κανείς είναι σαν τη Γερμανία μέσα σε μία μηχανή του χρόνου που μας μεταφέρει στο παρελθόν. Τώρα όμως είναι η ώρα να περάσουμε στο μέλλον, να επανέλθουμε στην κανονικότητα και αυτό θα πρέπει να το πετύχουμε μόλις μας το επιστρέψει η κατάσταση της υγείας όλων μας να είμαστε και ειλικρινεί. Θα είναι δύσκολο να επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Δεν έχουμε λύσει και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι θα είναι δύσκολη η όλη διαδικασία. Θα είναι δύσκολε οι αποφάσει που καλούνται να πάρουν τα κράτη-μέλη και παρά τα περιθώρια ελιγμού που υπάρχουν. Γιατί κανεί δεν θέλει φυσικά ένα δεύτερο κύμα μολύνσεων. Και προφανώ όλοι παράλληλα ανησυχούν για την οικονομία και για τι συνέπειε που θα έχει ο COVID. Πράχει πρόθεσμα. Στο άμεσο μέλλον θα πρέπει να ξεκινήσει να κινείται και πάλι η Ευρώπη. Να σεβαστούμε βέβαια παράλληλα και τους κανόνες κοινωνικής ε, απόστασης. Μακροπρόθεσμα θα πρέπει να εμβαθύνουμε και να διευρύνουμε την, το Σέγγεν. Την επόμενη εβδομάδα θα εκδώσουμε την πρώτη κατευθυντήρια γραμμή για την άρση των ε, περιορισμών και σε ό,τι αφορά και τον κλάδο του τουρισμού. Εδώ είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Τα κράτη-μέλη εισήγαγαν διαφορετικά μέτρα και μάλιστα με μη συντονισμένο τρόπο. Το πώ αυτές οι εθνικοί περιορισμοί θα μειωθούν θα είναι δύσκολο, θα πάρει χρόνο. Μπορούμε να το πετύχουμε όμω. και θα προτείνουμε μια βαθμιαία προσέγγιση για την άρση των συνοριακών ελέγχων. Η άρση των περιορισμών αυτών μπορεί να βασιστεί σε κάποιους σαφεί δείκτε για την διάδοση του ιού και για την κατάσταση του υγειονομικού συστήματο. και σε ό,τι αφορά τα μέτρα κοινωνικής απόστασης και άλλα προστατευτικά μέτρα. Τώρα λοιπόν, εξετάζουμε τρία βασικά ζητήματα. Καταρχάς, τις βασικές, ε, τους βασικούς όρους για την άρση συνοριακών ελέγχων, κατά δεύτερον μια συντονισμένη προσέγγιση και κατά τρίτον τι υποστήριξη, τι καθοδήγηση αναμένουν και χρειάζονται τα κράτη-μέλη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ό,τι και να κάνουμε, οι περιορισμοί αυτοί θα αρθούν βάσει των αξιών μα. Δεν θα υπάρξουν διακριτική μεταχείριση. Τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να ανοίγουν ε, ε, τα σύνορά του για πολίτε από κάποια χώρα και όχι για κάποια άλλη χώρα. Αυτό είναι βασικό μακροπρόθεσμα. Θα πρέπει να πετύχουμε κάτι, κάτι παραπάνω από την επιστροφή στο status Θα πρέπει να ενισχύσουμε το Σέγγεν και το νομικό του υπόβαθρο, να προετοιμαστούμε για τις προκλήσεις του σήμερα, του αύριο. Όταν πέντε κρατημέλη υπέγραψαν τη συνθήκη του Σέγγεν το 1995, δεν είχε πέσει το τείχος και δεν, είχε, δεν υπήρχε το ίντερνετ. Τώρα ξέρουμε πώ έχουν προχωρήσει τα πράγματα. Καταρχάς, θα ήθελα η Ρουμανία, η Κροατία και η Βουλγαρία να μπουν στο Σέγγεν. Μία καλή λοιπόν ζώνη Σέγγεν θα εξαρτηθεί από τη σωστή εφαρμογή του κεκτημένου του Σέγγεν. Γιατί ένα πρόβλημα σε ένα κράτο μέλο θα έχει συνέπειε σε όλε τι υπόλοιπε χώρε και θα θέσει σε κίνδυνο το Σέγγεν. Για να υπάρξει μεγαλύτερη λοιπόν, εμπιστοσύνη θα πρέπει να ε, μαθαίνουμε και τις σχέσεις μας με τρίτες χώρες. Με μια πιο βαθιά και συντονισμένη ζώνη Σέγγεν θα πρέπει να χρειαστεί και μια καλύτερη πολιτική θεωρήσεων. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τους ε, κατοίκους τρίτων χωρών σε ό,τι αφορά την σταδιακή άρση των μέτρων. Αυτό θα ε, έχει επίδραση και στους τομείς του τουρισμού. Χρειάζεται λοιπόν μια κοινή προσέγγιση για τη μετανάστευση και αυτό θα κατοχυρωθεί στο επερχόμενο σύμφωνο. Και κατά τρίτον φυσικά το θέμα της ιστορικής ασφάλειας, γιατί μια ισχυρή ευρωπαϊκή ε, προσέγγιση για την καταπολέμηση ε, του εγκλήματος και του ψηφιακού, της ψηφιακής απάτης θα σημαίνει ένα ενισχυμένο πληροφοριακό σύστημα. Προτιμάζω λοιπόν προτάσεις για την ενίσχυση του Σέγγεν, καταρχάς για πιο σωστή εφαρμογή. Ε, Εναλλακτικέ λοιπόν για τους συνοριακούς ελέγχους, για παράδειγμα από την αστυνομία, διαστοριακή συνεργασία, ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου. Για να προωθηθεί επίσης η εμπιστοσύνη ανταλλαγή ε, πρακτικών λύσεων και πρωτοβολιών. Για παράδειγμα, ένα ανανεωμένο διάλογο ε, με όλα τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά το καθεστώ του Σέγγεν. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να εξασφαλίζουμε ότι το νομικό πλαίσιο του Σέγγεν αρμόζει για την αντιμετώπιση των τρέχουσων προκλήσεων και των μελλοντικών προκλήσεων. Είμαστε λοιπόν λίγε μέρε πριν από την ημέρα τη Ευρώπη. Να μην ξεχνάμε από τη διακήρυξη του Σούμαν πριν από 70 χρόνια και το παραθέτω η Ευρώπη δεν θα οικοδομηθεί με μιας με βάση ενός σχεδίου. Θα πρέπει να υπάρξουν αλληλεγγύη σε πολλούς τομείς και νομίζω ότι αυτό ισχύει και για την ανάκαμψη μετά από αυτή τη σοβαρή κρίση μέσα στην οποία βρισκόμαστε ακόμα τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Λέει η κυρία Παγκάθα. Ακριβώς όπως είπε ο πρόεδρος, τώρα θα αρχίσει ο γύρος τραπέζι με τις ερωτήσεις των συντονισμών. Έχετε μαξιμου τρία λεπτά, ακριβώς όπως ε, είπε εκείνος. Και τώρα η κυρία Μετσόλα για το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ Επίτροπε που ήρθατε. Πλησιάζει το Καλό και έχουμε το ρόλο σε όλα αυτά τα σκάφη που βυθίζονται ε, γεμάτα μετανάστες και τα κρατημέλη για άλλη μια φορά πασχίζουν να βρουν κάποιες ε, προσωρινές λύσεις και θεωρούμε ότι είναι εφικτό να υπάρξει συμφωνία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει ενιαία ε, στάση και έτσι να λύσει αυτά τα προβλήματα, να τα αντιμετωπίσει και να μην πάσχει του κάθε κράτο μόνο το Εδώ και καιρό λέμε ότι χρειάζεται να υπάρξει κατανομή τη ευθύνη. Το ΕΛΚ θεωρεί ότι αυτό θα πρέπει να γίνει με κάποιο είδου ε, έκφραση αλληλεγγύη που να έχει κάποιο νόημα και να υπάρχει και ένα καινούριο πλαίσιο για την μετεγκατάσταση και θεωρούμε ότι όλα τα κρατημέρια θα πρέπει από κοινού να έχουν την ευθύνη και από ό,τι είπαμε να αντιμετωπίσουμε ε, τους λάθρους διακινητές, όλους αυτούς που εκμεταλλεύονται τον κόσμο για να κερδίσουν. Δεν θα πρέπει να πνίγεται ο κόσμος, θα πρέπει να έχουμε ασφαλείς λιμένες σε όλες τις ακτές της Μεσογείου και εκεί να υπάρχει ασφαλής ε, αποβίβαση και οπότε και αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ομαδικά. Οπότε επίσης να θωρακίζουμε τα σύνορα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη των 10.000 συνοφυλάκων και κάτι να κάνουμε για όλους αυτούς οι οποίοι δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για προστασία, να πάνε πίσω στις χώρες τους, αλλά να είναι σεβαστά τα δικαιώματά τους, να χρησιμοποιήσουμε ό,τι μέσα έχουμε, ώστε να υπάρχει συνεργασία με τις χώρες εκείνες και θα πρέπει αυτοί να δεχτούν τους πολίτες τους πίσω. Επίσης, να επενδύσουμε περισσότερα στις σχέσεις με τις τρίτες χώρες, αυτό σημαίνει περισσότερα χρήματα, πιο ευφυείς πρωτοβουλίες και να αναπτύξουμε ό,τι οι σχέσει χρειάζονται για να υπάρξει συνεργασία για την μετανάστευση. Θεωρούμε ότι μπορεί να είναι πρωτοπόρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπράβο, κυρία Επίτροπε, καλά τα είπατε νομίζω ότι υπάρχουν θερμιντικέ ε, ακτίνε ε, ελπίδα από τα κράτη-μέλη και αυτού που ήταν στην αρχή πιο διστακτικοί. Αλλά το θέμα είναι τελικά πώ θα μπορούσαμε να απεμπλέξουμε την κατάσταση από το σημερινό διέξοδο, γιατί έχουμε φτάσει σε κρίσιμο σημείο ίσως ε, ε, όσο πιο κρίσιμο ε, έχει ποτέ συμβεί και θα πρέπει μένως όλοι κάτι να κάνουν. Η Μαΐτα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τους σοσιαλδημοκράτες, η κυρία Ζίπελ. Η σύνδεσή σας είναι καλά. Ζίπελ. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ πάρα πολύ και την Επίτροπο Γιώχανσον. Και υπογραμμίζω αυτά που είπατε εισαγωγικά για το θέμα της ασφάλειας. Όντω, οι εγκληματίε προσαρμόστηκαν πάρα πολύ εύκολα και σε ό,τι αφορά την απάτη με τα φάρμακα, την προστατευτικό εξοπλισμό, αλλά και σε ό,τι αφορά τι απάτε για την απόσπαση ε, χρημάτων από ε, επιχειρήσει. Και το θέμα τη ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών, κατά των παιδιών, είναι ένα θέμα το οποίο δυστυχώ μα απασχολεί έντονα. Ευχαριστώ ιδιαίτερα λοιπόν για το γεγονό ότι παρουσιάσατε ε, το τι διαπροσωπικές σχέσεις υπάρχουν σε διασυνοριακό επίπεδο στην Ευρώπη και παρά το γεγονός ότι στην αρχή υπήρχαν μαζικοί, μαζικός έλεγχος και κλείσιμο των συνόρων, κατέστη σαφές παρά, παρά όλα αυτά πόσο σημαντικό είναι, πόσο σημαντική είναι η ζώνη Σέγγεν για το θέμα τη μετανάστευση και του ασύλου. Κυρία Επίτροπε, είπατε ότι έχουμε 1.600 ασυνόδευτου ανηλίκου οι οποίοι θα απορροφηθούν από τα κράτη-μέλη. Δυστυχώ, εγώ διαπιστώνω ότι εδώ στα κράτη-μέλη υπάρχει ε, μια πολύ επιλεκτική προσέγγιση. Λέμε ότι ναι, θα δεχτούμε κάποιους ε, ανηλίκους, αλλά μέχρι 14 ετών, μόνο κορίτσια και βλέπω συνολικά μια πολύ περιορισμένη κίνηση, γιατί είναι τεράστια αυτή η ανθρωπιστική δράση. Θα πρέπει να συμπεριληφθούν και νέοι οι οποίοι ε, έχουν ε, προβλήματα. Είναι παράλογη η κατάσταση. Από την άλλη, η κυρία Φοντερ Λάιεν ε, πριν από την εκλογή τη είχε ανακοινώσει ένα νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση. Αναρωτιέμαι, διαρωτώ με, τι θα είναι καινούριο αυτό το σύμφωνο τελικά. Καινούριο ο τίτλο. Και θα είναι ίδιο το περιεχόμενο. Αισθητική φύση θα είναι οι αλλαγέ. Έχω κάποιε συγκεκριμένε ερωτήσει να κάνω το νέο σύμφωνο όντω θα αλλάξει και θα έχει ω συνέπεια τη μετατροπή του Δουβλίνου. Θα υπάρξουν μετακαταστάσει, θα υπάρξουν ε, βιώσιμη ε, διαχείριση των μεταναστευτικών ορών, θα υπάρξουν κυρώσει άμα δεν τηρηθούν οι διδάξεις. Και τι γίνεται με την εκένωση των ε, καταβλισμών στα ελληνικά νησιά με την μετεγκαταστασή τους στην υπηρετική χώρα. Πόσο έχουν προχωρήσει όλα αυτά. Και μία τελευταία, τελευταία ερώτηση. Η κυρία Φοντερ ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει αυτό το νέο σύμφωνο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σύνολό τη τι α, ε, σκοπό έχει να κάνει για να πετύχει να σημειωθεί κίνηση στα κρατημέλη και επιτέλους να έχουμε ένα πακέτο ασύλου με αλληλεγγύη, στο οποίο να συμμετέχουν όλα τα κρατημέλη και το οποίο θα διασφαλίζει τα βασικά δικαιώματα, τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων μας. Ε, una... Σας ευχαριστούμε, λέει η Πρόεδρος, και τώρα κάτι θέλω να σας πω σε όλου σε όσους ε, ψηφίζουν. Από ό,τι μου λένε από την γραμματεία, μέχρι τις 3 μπορείτε να ψηφίσετε. Μέχρι τότε είναι ανοιχτή η ψηφοφορία. Άρα μέχρι τις 3. Επομένως έχετε ακόμα λίγη ώρα. Πάμε τώρα. Η συντονίστρια από το Ρήνιο, κυρία Ινετφέλτ. Μας ακούτε? Ναι, σας ακούω, λέει η κυρία Ινετφέλτ. Ελπίζω ότι και εσείς μπορείτε να μας ε, ακούσετε καθαρά. Κυρία Επίτροπε, σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Και πάλι ευχαριστούμε γιατί έρχεστε τακτικά να μας δείτε και καταβάλλετε προσπάθειες σημαντικές προς τη σωστή κατεύθυνση και θα ήθελα πρώτα-πρώτα να πω το ότι όταν βλέπουμε τι γίνεται στη Μεσόγειο, στα νησιά τα ελληνικά, από τη Λιβύη έρχεται κόσμος προς Μάλτα και Ιταλία και διάφορα άλλα τα οποία συμβαίνουν διαπιστώνω ότι κάποια κράτη-μέλη δεν υποστηρίζουν τους υπολείπους. Αυτό είναι μεγάλη ντροπή. Και η λέξη κλειδί εδώ είναι αλληλεγγύη. Όλοι την επικαλούνται. Τώρα που κάποιες χώρες, κάποια κόμματα λένε ότι είναι πρωτοπόροι για τα ανθρώπινα δικαιώματα, της αξίες, όμως στην πραγματικότητα γράφουν στα παλιά τους υποδήματα όλες αυτές τις προσπάθειες που γίνονται. Και λυπάμαι γιατί ούτε η δική μου χώρα ε, δεν δείχνει όση ελεγγύη θα ήθελα. Τώρα, μπορείτε να μας πείτε δυο λόγια παραπάνω όσον αφορά το τι ισχύει για το σύμφωνο μετανάστευση, γιατί ακούγονται διάφορα όσον αφορά την υποστήριξη, η έλλειψη υποστήριξης, ιδίω όσον αφορά την νόμιμη μετανάστευση. Και σε άλλε συναντήσει είχατε πει ότι δεν θα υπάρξει νομοθεσία για την ε, νόμιμη μετανάστευση. Ίσως αργότερα κάποιες με απλώς συντονιστικό χαρακτήρα. Η υποτική μα ομάδα θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντική ε, αυτή η υπόθεση τη νόμιμη μετανάστευση και θέλουμε να μπει στο νομοθετικό πακέτο. Επίσης, τι γίνεται όσον αφορά τι επαναπροωθήσει και αποθήσεις από τη Μάλτα. Τους στέλνουν πάνω σε ψαροκάικα πίσω στη Λιβύη το ερευνάτε, μπορείτε να μας επιβεβαιώσετε ότι τα ξέρει αυτά η Frontex. Τρίτο και τελευταίο, διαπιστώνεται ότι τα μέτρα καταπολέμησης της επιδημίας γνωρίζουν μια πολύ μεγάλη ποικιλία χώρα και αυτό έχει σχέση και με την μετανάστευση. Πώς να πάνε οι μετανάστες να ζητήσουν άσυλο ή να βρουν δουλειά ε, να κάνουν. Κάποιες χώρες ε, είναι πιο ρεαλιστικές, πιο ευμενείς όσον αφορά την αντιμετώπιση αυτών των ανθρώπων, άλλες δίνουν ή δεν δίνουν, άλλες άσυλο. Εσείς προβαίνετε σε συστάσεις με τις χώρες που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους. Ευχαριστούμε, λέει πρόεδρος, για το ID. Άννα Λίζα Ταρντίνο. Μας ακούτε? Κυρία Ταρντίνο. Sí. Vamos a... Ας περιμένουμε λίγο, διότι από ό,τι φαίνεται θα καταστεί εφικτή η σύνδεση με την κυρία Ταρντίνο. Usted pulsar... Πρέπει να πατήσετε το κουμπί, κυρία Ταρντίνο. Πατήστε το κουμπί. Bien. Α, ωραία. Η κυρία Ταρντίνο. Πολύ ωραία, έχετε το λόγο. Ναι, ναι, είμαι συνδεδεμένη τώρα νομίζω. Με ακούτε? Ναι, ναι, ναι, σας ακούμε λέει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Εγώ θα ήθελα να σταθώ σε αυτό που είπατε για τα πρόσφατα της Europol της 34ου. Τότε είπαμε ότι θα πρέπει να καταγραφεί η σχέση COVID και οργανωμένου εγκλήματος. Είπαμε ότι υπάρχει εκθετική αύξηση, το είπατε κι εσείς, του Ιντερνετικού εγκλήματος. Τι γίνεται όσον αφορά επίσης την απομίμηση, την παραποίηση φαρμάκων και προστατευτικού υλικού, γιατί κυκλοφορούν πάρα πολλά τέτοια μη πιστοποιημένα. Και επίσης όσον αφορά ε, κάποια δίθεν εμβόλια διαπράστονται απάτες. Οπότε θα πρέπει να υπάρξει κάποιο στρατηγικό σχέδιο και θα πρέπει επίσης να αναβαθμίσουμε τελωνιακούς και συνοριακούς ελέγχους τα εξωτερικά σύνορα και να δούμε τι θα γίνει με τις αρμοδιότητες Frontex, να υπάρχουν διαδικασίες πιο αυστηρές και έτσι να διώκονται οι παράνομοι και να προστατεύονται οι καταναλωτές και η υγεία τους. Και τώρα για να δούμε τι γίνεται όσον αφορά τους μετανάστες και να επανέλθουμε στα όσα ισχύουν τις αφήξεις λάθρων μεταναστών οι οποίοι ε, έρχονται όλο ένα και περισσότεροι από τη μία βδομάδα στην άλλη και αυτό γίνεται ε, με συνενοχή και ευθύνη της τελικής κυβέρνησης. Έχουμε αύξηση 400% σε σχέση με πέρσι στην ε, η Ιταλία επίσης ε, έρχονται και κυκλοφορούν ελεύθερα γιατί δεν υπάρχει κάποιο είδους τρόπος τακτοποίησης του θέματος. Άρα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι λαθροδιακινητές, ε, αυτοί που κερδίζουν για αυτά τα οποία κάνουν. Να δούμε το ότι επίσης έχει πληγεί η αφρικανική οικονομία. Ε, και αυτό θα συμβάλλει στη λαθρομετανάστευση. Θα πρέπει βέβαια να μπορέσουμε να επιστρατεύσουμε κάποιους μετανάστες οι οποίοι θα έχουν χαμηλό κόστος. Έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες λαθρομεταναστών. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με αυτούς που έχουν γεμίσει ε, την Ήπεθρο και αυτοί θα καταστούν τελικά όσον αφορά την γεωργία θα γίνουν δούλοι και έτσι θα πρέπει να δοθούν κάποια, να γίνει κάποια προσπάθεια για να μην έχουν κίνητρο ελαφρομετανάστες. Οπότε παρακαλώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σταματήσει αυτό το δουλεμπόριο ε, που τελικά καταλήγει στην πατρίδα μας. Σας ευχαριστούμε εμείς για τους πρασίνους. Στρίκ, κυρία Στρίκ. Μας ακούτε. Sí, señora Strick. Yes. Bien, <laughs> le escucho. ¿Tiene ακούμε, σας ακούμε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και την κυρία Γιώχανσον για τη δέσμευσή της για να υπάρξει μεγαλύτερη εναρμόνιση και πιο πολύ αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών. Όπω ξέρετε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέμεινε στην βελτίωση τη κατάσταση και των όρων διαβίωση σε ό,τι αφορά τους τούντε, άσυλο στα ελληνικά νησιά και επίσης επιμείναμε στα μέτρα προληπτικής εκένωσης για να προστατευτούν κατά του ιού. Αυτό ακόμα δεν έχει γίνει. Δεν έχει γίνει σε, μεγάλο, σε μεγάλη κλίμακα τουλάχιστον η κατάσταση επιδεινώνεται με πυρκαγιές στη Σάμο. Έλλειψη βασικών υπηρεσιών που είναι απαραίτητες. Η Επίτροπος λοιπόν μπορεί να μας εξηγήσει τι είδους μέτρα λαμβάνονται στην παρούσα φάση για να βελτιωθεί η κατάσταση. Επίσης, πώς εκτιμά τους νέους νόμους που βρίσκονται υπό συζήτηση στην Ελληνική Βουλή. Γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν θέματα ακόμα. Ακόμα περιμένουμε την υλοποίηση του προηγούμενου νομοσχεδίου της Ελλάδας. Μπορείτε λοιπόν να μας δώσετε μια εκτίμηση σε ό,τι αφορά τα διατάγματα της Ελλάδας και τα, τους νόμους. Δεν μπορεί φυσικά η Ελλάδα να τα πετύχει όλα αυτά μόνη της. Χρειάζεται πολύ, πιο πολύ αλληλεγγύη για την ε, μετεγκατάσταση, για την ανάληψη κοινών ευθυνών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς εκτιμά τη στάση των κρατών μελών. Διαβλέπει δυνατότητε να ενισχυθεί η αλληλεγγύη. Και τι λέει αυτή η στάση για τις νέες προτάσεις του συμφώνου. Πώς μπορούμε να δώσουμε ε, εξασφάλιση, πώς μπορούμε να δώσουμε δικλείδες ασφαλείας για την ανάλεψη ευθυνών. Και σε ό,τι αφορά την κατάργηση επίσης ε, της διατάξης για την ευθύνη του πρώτου κράτους εισόδου. Το θέμα φυσικά δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Κοιτάμε και την διακήρυξη της Μάλτας και διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει υποστήριξη από κάποια κράτη-μέλη. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει ε, με την κατάσταση μετά την ε, απόβαση των ανθρώπων αυτών. Αυτό έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο. Η Επίτροπος λοιπόν μπορεί να τα επιβεβαιώσει όλα αυτά. Και τι κάνει για να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Επίσης ακούμε για επαναπροωθήσεις και με πάσα σαφήνεια από πλευράς της Μάλτας υπάρχει ομολογία σε ό,τι αφορά τη συνενοχή αυτή από την κυβέρνηση της ε, Μάλτας. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε λοιπόν αυτό τι θα σημαίνει, τι παράδειγμα θα δώσει και σε άλλα κράτη-μέλη. Τι θα κάνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι έκανε και η Frontex. Εκείνη το Σαββατοκύριακο του Πάσχα η ακτοφυλακή της Λιβύης έκανε διάφορες ε, δράσεις διάσωσης. Ε, ήταν ενήμερη η Frontex, ήταν ενήμερη η Frontex για το τι συνέβαινε ε, στα σύνορα της Μάλτας. Ενημερώστε μας. Και επίσης, ξέρουμε ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης στα σύνορα της Λιβύης δεν είναι ασφαλείς και επίσης γνωρίζουμε ότι η κατάσταση για τους μετανάστες στη Λιβύη είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Άρα, αυτό τι σημαίνει για την συνεχιζόμενη συνεργασία με την Λιβύη και την ακτοφυλακή αυτής. Ανησυχούμε. Αλλά έχουμε επιχειρήσει οι οποίε ε, ενισχύουν ουσιαστικά τη συνεργασία με την ε, ακτοφυλακή της Λιβύης. Υπάρχει επίσης ε, και παρακολούθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς επιτηρούμε την τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και πώς ε, εκτιμούμε την ε, μεταχείριση των μεταναστών. Ευχαριστώ. Για το ECR τώρα θα λάβει το λόγο ο Νικόλα Προκατσίνη. Μας ακούτε? Παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Ναι, με ακούτε, λέει ο κύριος Προκατσίν. Καλησπέρα σε όλους. Πρώτα-πρώτα Επίτροπε Γιωχάνσον, πρώτη ερώτηση. Οι τρομοκρατικές συμμορίες εκμεταλλεύονται αυτή την πανδημία για να βγουν μπροστά και να προβληθούν όπως ξέρουμε ότι έγινε και με το Ισλαμικό κράτος. Προσπαθούν μέσω της ε, προδημίας να προβάλλουν τις θέσεις τους και έτσι να διαδώσουν την Ισλαμιστική προπαγάνδα. Έχουμε το μηχανισμό τόσο ώστε να φρενάρουμε με τέτοιες δραστηριότητες. Επίσης θα πρέπει ταχαίως να εγκριθεί ο κανονισμός όσον αφορά την τρομοκρατία ως περιεχόμενο του ίντερνετ. Άρα θα πρέπει να κάνουμε περισσότερο για να καταβολήσουμε τέτοια προπαγάνδα. Δεύτερη ερώτηση. Μιλήσαμε για την έκθεση της ε, Europol. Τότε που αναφερθεί ότι υπάρχει διακίνηση λαθρομεταναστών κατά τη διάρκεια της επιδημίας. Και αυτό βέβαια επιβαρύνει υγειονομικά και οικονομικά τις ε, χώρες τις οποίες διαβαίνουν αυτοί οι μεταναστές. Οπότε, για πέστε μας, τι λέτε για αυτή τη διακίνηση των μεταναστών; Η ΜΚΟ θα αναλάβουν το πήγαινε έλα στην Λιβύη και έτσι να πέφτουν στην αγκαλιά των λαθροδιακινητών ή μετανάστες. Αυτό δεν είναι λύση. Τι λέτε για το μεταναστευτικό γενικώ, δεν νομίζετε ότι τώρα η υγειονομική κρίση το θέμα το έχει παροξύνει και έχει κάνει ακόμα χειρότερη την κατάσταση με το μεταναστευτικό. Δεν πρέπει να είμαστε αφελείς νομίζω κύριε Επίτροπε ότι και το θέμα της μετεγκατάστασης αλλά και το θέμα των επαναπατρισμών είναι δύο λύσεις που έχουν αποτύχει. Άρα, επιτέλους, θα πρέπει να βρεθεί ο τρίτος δρόμος. Να δούμε πώς θα φρενάρουμε τις αναχωρήσεις. Θα πρέπει να γίνει διαχείριση αυτών των αναχωρήσεων. Να μπορέσουμε να φιλτράρουμε από εκεί ποιος δικαιούται και ποιος όχι την διεθνή προστασία. Θα πρέπει να είναι παρούσα, πολύ παρούσα η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά της οργάνωσης στη Λιβύη και σε όλα τα κράτη από όπου προέρχονται οι μεταναστές. Μόνο έτσι μπορέσουμε να κάνουμε κάτι και να ανακουφιστούν οι χώρες όπως η Ιταλία, Ισπανία, Μάλτα που θα πρέπει πέραν του υγειονομικού να αντιμετωπίσουν τώρα και το μεταναστευτικό. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Για την Ιγκούε. Κυρία Γιώργ, κύριε Μπιόρκ. Με είδατε, με είδατε. Ναι, ναι, ναι. Εδώ είμαι. Έχετε το λόγο. Δεν σας βλέπουμε όμως. Απλώς σας ακούμε. Τώρα με ακούτε, όχι λέει ο πρόεδρος. Can you hear me now? Τώρα, με ακούτε. Σα ακούμε, σα ακούμε, επαναλαμβάνει πρόεδρος. Δεν σα βλέπουμε. Να, μάλιστα, τώρα σα βλέπουμε. Έχετε το... Okay. So, I will try... Να προσπαθήσω. Και πάλι. Σας ευχαριστώ λοιπόν που παρευρεθήκατε στην ψηφιακή αυτή τηλεδιάσκεψή μας. Είναι πολύ χρήσιμη αυτή η ανταλλαγή απόψεων. Τρία πράγματα θέλω να πω και κάποια τα ακούσαμε ήδη από τους συναδέλφους. Θα τα αναφέρω εντάχει. Το θέμα λοιπόν το πρόμα, το θέμα της, α, ε, α, των ελληνικών νησιών. Όπως ξέρετε, η άποψή μας είναι ότι έχουν γίνει πολύ λίγα και πολύ αργά. Και το να μένουν στις φυλακές ε, ή αιτούντες άσυλο ε, στα νησιά ε, δεν είναι τμήμα της λύσης. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Χρειάζεται επανεγκατάσταση. Αυτή είναι η λύση. Αυτή θα πρέπει να είναι η λύση. Ακόμα και σε τέτοιες δύσκολες περιόδους. Ήταν 6.000 τα άτομα αυτά και είχα πάει τότε να επισκεφθώ και ήδη ήταν υπερβολικά γεμάτο. Δεν τολμώ καν να φανταστώ τι γίνεται σήμερα. Τονίζω λοιπόν αυτή το είναι έκκληση για μετεγκατάσταση. Δεν υπάρχει οποιοδήποτε εμπόδιο για την μετεγκατάσταση από τα νησιά. Τι κάνετε λοιπόν, ρωτώ, για να το πετύχετε αυτό, για να προχωρήσει το μέτρο αυτό της ε, επανεγκατάστασης, της μετεγκατάστασης σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεύτερη ερώτηση σε ό,τι αφορά την επαναπροώθηση. Το έθεσαν κάποιοι συνάδελφοι. Εγώ έχω δει με τα αιτία μου τα μάτια στην Κροατία επαναπροωθήσεις στα σύνορα με τη Βοσνία Τι γίνεται λοιπόν εκεί Έχω δει εικόνες από ανθρώπους που όχι μόνο τους ληστεύουν, όχι μόνο τους χτυπούν, αλλά τους ψεκάζουν. Τι κάνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να σταματήσουν αυτές οι επαναπροωθήσεις. Από την Κροατία στη Βοσνία Ζεγοβίνη και στα θέματα αυτά της ε, επαναπρόθεση προ Ανατολά ε, από τη Μάλτα. Θα πρέπει να συζητηθεί αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τρίτη ερώτηση. Για τα θέματα διάσωση και αναζήτησης. Εδώ η κατάσταση την έτησε και ο συνάδελφος προηγουμένως. Βλέπουμε λοιπόν ανθρώπους και σκάφη τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και τα οποία τα αφήνουμε με επιμέρειες στην τύχη τους. Τι γίνεται λοιπόν από τη Frontex. Χρειάζεται αλληλεγγύη. Να υπάρξει κατάσταση των ατόμων αυτών που χρειάζονται ένα ασφαλές περιβάλλον. Τι κάνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αντιμετωπίσει αυτή την επωνίδιστη κατάσταση σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάποιες περιπτώσεις δεν σηκώνουν καν τηλέφωνο. Είναι ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να στραφεί προς την Frontex και να ζητήσει διευκρινήσεις για το τι κάνουν. Δεν βοηθούν τους μετανάστες και βάζουν σε κίνδυνο, συγκεκριμένο κίνδυνο τη ζωή των ανθρώπων. Ρωτώ λοιπόν τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προ την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, πρόεδρο. Πρόεδρος. Κύριε Λόπεθ Αγγιλάρ, κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Μα ακούτε? Έχετε καλή σύνδεση? Ναι, ναι. Ναι, ναι, και μπόρεσα να τα ακούσω όλα. Και ευχαριστώ βεβαίω και την Επίτροπο να σας πω ποιες ε, ανησυχίες υπάρχουν, τι προέκυψε από ψηφίσματα, από ψηφοφορίες σε σχέση με αυτά τα οποία έχει θίξει η Επίτροπος και ο κύριος Μπαρόσο επίσης τα έχει πει η συνθήκη του Σέγγεν είναι από τα πιο πολύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τώρα μας λείπει. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που γίνεται αναστολή ε, της καταργήσεως των εσωτερικών συνόρων και έτσι να υπάρχει ορισμός των φυσικών προσώπων. Είχαμε το 15, το προσφυγικό, 15 με 16 και τότε είχαμε έγκυρη αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπήρξε μια ανακοίνωση που υπενθύμησε στα κράτη-μέλη ότι ακόμα και υπό δύσκολε συνθήκες ακόμα και όταν έχουμε κάποια μονομερή μέτρα κάποιων κρατών μελών ακόμη υπάρχει δίκαιο υπάρχουν δεσμευτικέ διατάξεις για όλους και αυτό καλύπτει και τον κώδικα Σέγγεν 28, 29 και 30 άρθρα του κώδικα Σέγγεν. Εκεί διατυπώνεται ρητό ότι θα πρέπει να λάβουν τα κράτη-μέλη μέτρα τα οποία να έχουν συγκεκριμένη διάρκεια και οριζόντια ε, οριζόντιο χαρακτήρα συντονισμού και να έχουν κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να υπάρχουν εγγύησεις για την τήρηση του κοινοτικού δικαίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι ο φύλακας των συνθήκων. Τι θα γίνει κύριε Επίτροπε, πώς θα μπορέσουμε σύντομα να υπάρξει επιστροφή στην κανονικότητα του Σέγγεν. Έστω και βαθμία να υπάρχει ελεύθερη διακίνηση γιατί αυτό είναι σημαντικό και για την οικονομική ανάκαμψη αλλά και για την επιβίωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και επιμένω ότι είναι πολύ σημαντική πράσινη διάδρομη για τους εποχιακούς εργαζόμενους. Πολύ σημαντικό για τις επιχειρήσεις αλλά και για την γεωργία. Και αυτό αφορά όλη την Ένωση και όχι μόνο κάποια κράτη-μέλη. έχουμε το ψήφισμα του Απριλίου και το είπαμε στην παράγραφο 40 θα πρέπει να υπάρχουν πράσινοι διάδρομοι όχι μόνο για την προμήθεια των βασικών αγαθών αλλά και για τους εποχιακούς. Αυτή είναι πολύ σημαντική όσον αφορά την επιβίωση της γεωργίας και αυτοί οι εποχιακοί θα πρέπει να μπορούν να περάσουν να φτάσουν εκεί που τους χρειάζονται τα κράτη-μέλη και η Γεωργία. Και επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο θέμα οικονομίας, είναι θέμα επιβίωσης του ιδιώδους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνδέεται με το Σέγγεν. Τώρα, για το άσυλο. Συμφωνώ με όλες τις ανησυχίες που διατυπώθηκαν και επαναλαμβάνω ότι έχουμε αυτά τα σκάφια προς Μάλτα, από τη Λιβύη, από την Αφρική προς τα Κανάρια. Πολύ ενσχυτική η κατάσταση. Θα πρέπει να υπάρξει ελεγγύη με δεσμευτικού κανόνες, πλαίσιο με την κατάσταση και ξέρετε για το πλαίσιο έρευνας και διάσωσης που δεν το περάσαμε για δύο ε, ψήφους. Εγώ ήμουν ο εισηγητής. Άρα κάντε κάτι να εξασφαλίσετε ότι στο καινούριο σύμφωνο θα υπάρξει ένα κεφάλαιο για ευρωπαϊκό α, ε, πλαίσιο έρευνας και διάσωσης. Να μην έχουμε εμβαλωματικά ε, μέτρα κατά, κατάτμιση του καθεστώτος που ισχύει, ο καθένας να κάνει ό,τι του έρχεται, να υπάρχει χαλασμένο τηλέφωνο στην ενόηση και επίσης για τους ανηλίκους που πρέπει να μετεγκατασταθούν. από τους καταβλισμούς που έχουν ξεχυλίσει τα ευρωπαϊκά νησιά. Θα πρέπει κάτι να γίνει. Αλλά τι γίνεται με τις οικογένειες αυτών των ανηλίκων, τι γίνεται με τις μανάδες τους, τι γίνεται με ε, τους ε, ασυνόδευτους. Ε, θα πρέπει να υπάρξει κάποιο είδους επανένωση. Βλέπουμε ότι κάποιοι ανήλικοι πάνε από τα νησιά στην υπηρετική χώρα στην Ελλάδα. Θα πρέπει όλα να γίνουν με αλληλεγγύη. Να κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε μια πολύ μακρύ κατάλογο αγορετών. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, πρόκειται περί εγκλημάτων ε, και γι' αυτό σας λέω ότι ανησυχούμε. Χρειάζεται μια εσωτερική στρατηγική, χρειάζεται μια επικαιροποιημένη προ... για όλα αυτά τα εγκλήματα που έχουν σχέση με τη διαχείριση της πανδημίας. Και σας ευχαριστώ. Εμείς, λέει ο Πρόεδρος, πριν αρχίσει ο πρώτος γύρος απαντήσεων της Επιτρόπου, θα πρέπει να υποβάλω ένα σύντομο ερώτημα. Αύριο όλοι θα θυμηθούμε τα θύματα που είναι πάνω από 30.000 Ευρωπαϊκοί στα θύματα της πανδημίας και ελπίζω και εμείς όπως οι προκαθήμενοι μας σε αυτές τις θέσεις να δείξουμε υπευθυνότητα. Πολλά ήταν τα ερωτήματα κύριε Επιτροπέ. Εγώ θέλω να σας πω κάτι όσον αφορά το πόσο ευάλωτοι είμαστε στο ηλεκτρονικό εμπόριο και ότι υπάρχει για το κυβερνό έγκλημα τώρα ατιμορρησία. Μας είπε η Επιτροπή ότι τέλη του έτους θα ολοκληρωθεί ε, η αναθεώρηση του AIDAS, του κανονισμού, για την ηλεκτρονική εξακρίβωση βάσει ε, κάποιες ταυτότητος να καταπολεμήσουμε το κυβερνό έγκλημα. Αυτό χρειάζεται, γιατί έχουμε πολύ βαριά εγκλήματα και επίσης ατιμορρησία σήμερα. Σήμερα την εποχή της πανδημίας γνωρίζουμε ότι κάποιες από τις συνέπειες πανδημίας θα τραβήξουν και στο μέλλον. Και σας ερωτώ κύριε Επιτροπέ, μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει κάποια προτεραιότητα σε αυτό το θέμα, γιατί πρόκειται για κάτι το οποίο φύγει ε, το ζήτημα της αντιμετώπισης του βαριών εγκλημάτων. Θα πρέπει κάτι να γίνει για τον σχετικό κανονισμό της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Είναι κάτι που επήγει. Θα μπορεί, πρέπει να το προωθήσετε αυτό και είναι σημαντικό αυτό να το βάλετε στο πακέτο, στη δέσμη αυτή μέτρων για το COVID. Έχετε το λόγο των πρώτων κυκλοπαντήσεων, κύριε Επίτροπε, πριν αρχίσουμε το δεύτερο κύκλο ερωτήσεων τους βουλευτές. Μας ακούτε? Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και για όλες τις ερωτήσεις που μου υποβάλατε και πέρα από τις ερωτήσεις και για τις απόψεις που μου παρουσιάσατε, να προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις. Καταρχάς, στην κυρία Μέτσολα, να πω ότι ναι, θα χρησιμοποιήσουμε ό,τι εργαλεία έχουμε στη διάθεσή μας για να βρούμε καλή σχέσεις. Σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση, αλλά και για άλλους σκοπούς, να υπάρχει καλή σχέση με τις τρίτες χώρες. Η κυρία Ιντφέλτ επίσης έθεσε το ερώτημα της νόμιμης μετανάστευσης και αυτό προφανώς αποτελεί ε, βασικό στοιχείο της εταιρική σχέση με τις τρίτες χώρες, το οποίο επίσης θα πρέπει να εξασφαλίσουμε. Θα πρέπει να υπάρχουν νόμιμες οδοί για την ε, έλευση του κόσμου αυτού, αλλά και για την ε, μετακατάσταση όσων χρειάζονται διεθνή προστασία. Ναι, λοιπόν. Η κυρία Μέτσολα επίσης έδωσε πολλές ε, σημαντικές επιτυχίες ε, και συμφωνώ απόλυτα ότι κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να έχει κοινή ευθύνη. Να έχει μέρος της ευθύνης. Αυτό θα είναι ε, τμήμα της νέας πρότασης του νέου συμφώνου που προετοιμάζουμε. Αναγνωρίζω επίσης ότι το ΕΛΚ πρόσφατα υπέβαλε ένα πρόγραμμα για τη μετανάστευση και το άσυλο και ένα τμήμα αυτό να έχει συμπεριληφθεί. Ακούσαμε το σημαντικό θέμα της, ε, των γυναικών και των παιδιών. Μ' ανησυχεί ιδιαίτερως λοιπόν αυτό. Έχουμε δει σχεδόν σε όλα τα κράτη-μέλη δραματική αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών και σε κάποιες περιπτώσεις κατά των παιδιών. Αυτό δεν είναι αρμοδιότητα ουσιαστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πρέπει να πω ότι ως φεμινίστρια, ως γυναίκα, ανησυχώ ιδιαίτερως για τα περιστατικά αυτά. Το θέμα των ασυνόδευτων ανηλίκων και της μετεγκατάστασης αυτών. Πώς ε, γίνεται η επιλογή και διαλέγουν πραγματικά τα κράτη-μέλη ποιου ασυνόδευτου ανηλίκους ε, θα δεχτούν. Έγινε κανένα διάλογο με τα κράτη-μέλη. Ξεκίνησαν κάποια κράτη-μέλη με κάποιε μη ρεαλιστικέ απόψει για το ποιου θέλουν να δεχτούν αλλά καταλήξαμε με μια πιο ευρεία ομάδα ατόμων για με την εγκατάσταση. Επίση, έγινε διάλογο, λέω, και στην κυρία Σίπελ και στον κύριο Λόπε Αγγιλάρ, όχι μόνο για του ε, ασυνόδευτου ανηλίκου, αλλά και για τι γυναίκε, για τι οικογένειε, συγγνώμη, με παιδιά άρρωστα, που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στι προσπάθειε με την εγκατάσταση. Το νέο σύμφωνο, το οποίο θα παρουσιάσουμε, ελπίζω σύντομα, δεν θα είναι μόνο ένα σύμφωνο για διακοσμητικές ε, αλλαγές. Θα περιλαμβάνει και καινούργιες προτάσεις, αλλά θα ληφθούν επίσης υπόψη, προφανώς, και όλα όσα έχουν γίνει ως τώρα, μεταξύ των οποίων και όσα έχει κάνει το Κοινοβούλιο. Δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Θα ληφθούν υπόψη, λοιπόν, όλα όσα έχουν γίνει. Η κυρία Σίπελ επίσης ρώτησε για το τι κάνω για να εξασφαλίσω ότι θα γίνει αποδεκτό αυτό το νέο σύμφωνο σε ό,τι αφορά τα κράτη-μέλη. Σε ό,τι αφορά πριν ε, μάλλον επιβληθούν οι προορισμοί στα σύνορα, ε, σκόπευα να επισκεφτώ όλα τα κράτη-μέλη, να κάνω και συζητήσεις ε, με τα κοινοβούλια, με την κοινωνία των πολιτών, της ΜΚΟ. Προσπάθησα λοιπόν να βρω ένα γόνιμο έδαφος για την νέα αυτή πρόταση. Προς την κυρία Εντφέλτ. Να πω ότι συμφωνώ με τις απόψεις σας και είναι σημαντικό όλα τα κρατημέλη να επιδείξουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους και σε ό,τι αφορά τους ασυνοδότε ανήλικου, αλλά περιμένουμε εδώ κάποια κρατημέλη πραγματικά να επιδείξουν έμπρακτη αλληλεγγύη. Η νόμιμη μετανάστευση προφανώ και αποτελεί ένα βασικό στοιχείο του νέου συμφώνου. Για μένα είναι σημαντικό να προστατεύσουμε τα σύνορά μας και να είμαστε πιο αποτελεσματικοί σε ό,τι αφορά την επιστροφή αυτών που δεν χρήζουν διεθνούς προστασίας. Αλλά εκ παραλλήλου θα πρέπει να είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε και τους άλλους που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω νόμιμων οδών μετανάστευσης. Αυτό είναι βασικό στοιχείο του πακέτου. Σε ό,τι αφορά τη Μάλτα, και εγώ είδα αυτό το ρεπορτάζ στα μέσα για τις επαναπροωθήσεις. Είδαμε και φρεχτή απώλεια ζωών. Αυτό πραγματικά είναι κάτι τρομακτικό. Και προφανώς είναι από τα βασικά καθήκοντά μας να σώζουμε ζωές. Αυτό με ανησυχεί, λοιπόν. Και προφανώς και περιμένω από τις αρχές της Μάλτας να ερευνήσουν το τι πραγματικά συνέβη στην προκειμένη περίπτωση σε ό,τι αφορά το ρόλο της Frontex. Η Frontex έχει αναλάβει την επιτηρήση. Ενημέρωση επίσης των αρχών διάσωσης και των κέντρων συντονισμών της Μάλτας όταν υπάρχουν περιστατικά σε τέτοιες περιπτώσεις. Επίσης, Ξέρουν ότι οι αρχές της ε, Λιβύης είχαν κάποιους περιορισμούς κάποιες μέρες λόγω του ιού. Τώρα όμως πλέον έχουν ε, ξαναξεκινήσει με την άσκηση των καθηκόντων τους. Η επιχειρήση τη διάσωση είναι εθνική αρμοδιότητα. Δεν είναι ουσιαστικά αρμοδιότητα τη Frontex. Υπάρχει ρόλος επιτήρησης για το κατά πόσον είναι ενημερωμένη στην περίπτωση αυτή σε ό,τι αφορά τις επαναπροωθήσεις. Δεν ε, είμαι σε θέση να σας απαντήσω. Δεν έχω τις σωστές πληροφορίες ή να δώσω απάντηση στην ερώτηση αυτή. Και συμφωνώ με την κυρία Ιντφέλτ ότι ήταν πολύ ενθαρρυντικό το γεγονό ότι είδαμε κάποια κρατημέλη να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίε σε ό,τι αφορά του μετανάστε, ε, του ετούντε άσυλο, σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασία. Ε, στη συμπερίληψή τους στην κοινωνία σε αυτή την ε, κρίση, την πανδημία. Επίσης, ρωτήσατε κατά πόσον παρακολουθούμε τι κάνουν τα κράτη-μέλη σε αυτή την φάση σε ό,τι αφορά το άσυλο και την μετανάστευση. Ναι, Προφανώς και τα παρακολουθούμε όλα αυτά και έχει εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώς θα πρέπει να δράσουμε για να ακολουθήσουμε το δίκαιο και να ακολουθήσουμε και αυτά που επιτάσσει η τήρηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θελομελιδών δικαιωμάτων προς την κυρία Ταρντίνο. Όπως είπατε, ήταν πάρα πολύ σημαντική αυτή η έκθεση της Europol για το οργανωμένο έγκλημα και θα επηρεάσει προφανώς και τις προτάσεις που θα υποβάλουμε για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Ζητήσατε να διευκρινίσουμε κατά πόσον η Frontex θα μπορούσε να έχει κάποιο ρόλο σε ό,τι αφορά τους τελωνιακού ελέγχου, αν κατάλαβα σωστά. Αυτό είναι εκτός της εντολής της Frontex. Εκεί δεν μπορούν να έχουν κάποιο ρόλο σε ό,τι αφορά τα τελωνιακά ζητήματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το trafficking, τη διακίνηση ανθρώπων και την καταπολέμηση αυτού. Είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό. Πρόκειται για το ένα από τα χειρότερα εγκλήματα τα οποία υπάρχουν. Οι διακινητές προφανώς και σχετίζονται με τις συμμορίες οργανωμένου εγκλήματος διακίνηση ανθρώπων και διακίνηση ναρκωτικών. Ανάλογα με τις αλλαγές που γίνονται είναι σημαντικό λοιπόν να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την καταπολέμηση του φαινομένου σε ό,τι αφορά τη διακίνηση και εδώ θεωρώ ότι θα πρέπει να καταβάλουμε πιο έντονε προσπάθειε. Και κάτι άλλο σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να αλλάξει η ηλικία, θεωρώ, για τα δακτυλικά αποτυπώματα των παιδιών από τα 6 χρόνια. Για όσους ζητούν θεώρηση ή είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Europol είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να μπορέσουμε να καταστρέψουμε αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο των διακινητών. Προς την κυρία Στρίκ, να πω το εξή. Η προληπτική εκένωση των ευάλωτων ομάδων από τους καταβλισμούς, και η κυρία Μπιόρκ το έθεσε το θέμα αυτό, είναι υπό εξέλιξη, όπως είπα και εισαγωγικά. Όλα αυτά γίνονται με τις ελληνικές αρχές και με τις οργανώσεις του ΟΗΕ, τη UNHCR, για τους πρόσφυγες. Χίλια άτομα λοιπόν έχουν εκενωθεί από τους καταβλισμού, 392 άτομα μετακινούνται αυτή την εβδομάδα και την επόμενη εβδομάδα θα μετακινηθούν άλλα 600 άτομα. Αυτά είναι τα αριθμητικά στοιχεία τα οποία μας επιβεβαίωσε και η οργανώση γιατροί χωρίς σύνορα. 2.000 άτομα είχε αναφέρει ότι λίγο πολύ θα πρέπει να φύγουν από τους καταβλισμούς για να προστατευτούν σε περίπτωση που θα υπήρχε ξέσπασμα του ιού. Ως τώρα δεν υπήρχε απώλεια ζώων από την πανδημία στην Ελλάδα μεταξύ των μεταναστών στους καταβλισμούς. Ελπίζουμε ότι με τη μετακίνηση των ανθρώπων αυτών και των ασυνόδευτων ανηλίκων και κάποιων οικογενειών με παιδιά και με την εθελούσια επιστροφή, η οποία βρίσκεται υπό εξέλιξη στα ελληνικά νησιά. Θα επιλύσουμε το θέμα. Σε ό,τι αφορά το νέο νόμο της Ελλάδος, ο οποίος ε, περνάει από το Κοινοβούλιο, είμαστε σε στενή επαφή με τις αρχές της Ελλάδος. Και ξέρουμε ότι είχαμε και κάποιες συνομιλίες χθες, αν δεν κάνω λάθος, με τον Έλληνα Υπουργό για το θέμα αυτό. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξουν ε, κάποιες τροποποίησεις για να υπάρχει τήρηση του ευρωπαϊκού δικαίου. Η αποστολή ειρήνη τώρα. Δεν είμαι ενημερή για την ε, αποστολή αυτή. Είναι στην ε, αρμοδιότητα του Ιωσήπ Μπορέλ. Ξέρω ότι έχουν κάποια προβλήματα σε ό,τι αφορά την ε, επιχείρηση αυτή, αλλά δεν είμαι απόλυτα ενήμερη. Δεν μπορώ να απαντήσω λοιπόν. Προς την κυρία Προστασίνη. Ναι, υπάρχουν τρομοκρατικές ομάδες οι οποίες εκμεταλλεύονται την πανδημία. Ακραίες, ε, ακραίες σχηματισμοί. Και βλέπουμε ότι online υπάρχει ριζοσπαστικοποίηση. Αυτή η ιστορία του κορονοϊού τη χάνει εκμετάλλευση για την ενίσχυση δικτύων ριζοσπαστικοποίησης και συμφωνώ μαζί σας ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει αυτή η συζήτηση για το τρομοκρατικό υλικό το οποίο βρίσκεται στο διαδικτύο. Είναι σημαντικό. Και για τους διακινητές κάντε κάποια ερωτήματα, τα απάντησα ήδη. Επίσης, σε ό,τι αφορά το διάλογο με τις τρίτες χώρες. Είναι σημαντικό να βοηθήσουμε τις τρίτες χώρες σε αυτή τη ε, διαδικασία με την πανδημία. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα βοηθά το υγειονομικό σύστημα της Λιβύης για να ανοίξει και για τους μετανάστες. Είναι σημαντικό οι μετανάστες που βρίσκονται στη Λιβύη να έχουν πρόσβαση ε, υγειονομική περιθάλψη. Και εδώ συνδράμει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρία Μπιόρκ, ρωτήσατε και για την εκκίνωση για των νησιών. Απάντησα, φέρω, στην ερώτηση αυτή. Σε ό,τι αφορά την Κροατία τώρα. Πρόσφατα απέστειλα μία επιστολή στο Κοινοβούλιο και στην κυρία Φαγιόν. Βρισκόμαστε σε φάση εκτίμησης ακόμα του σχετικού σχεδίου. Χρειαζόμαστε πιο ακριβείς πληροφορίες από την Κροατία σε ό,τι αφορά την επαναπροώθηση και προγραμματίζουμε μία επίσκεψη για παρακολούθηση, η οποία προφανώς και αναβλήθηκε τώρα λόγω του ιού, αλλά θα λάβει χώρα το σύντομο δυνατόν. ανάλογα και με την εξέλιξη του ιού. Είχαμε επαφέ και με τον ε, διαμεσολαβητή στην Κροατία την προηγούμενη εβδομάδα και μαζί με τις ε, κροατικές αρχές και τον διαμεσολαβητή στην Κροατία εξετάζουμε το πώς θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε τα σύνορα της Κροατίας με πιο ενισχυμένο τρόπο θα πρέπει να ακολουθηθεί η αρχή της μη επαναπροώθησης, αλλά όλα αυτά θα αναφερθούν στην επιστολή. Η κυρία Μπιόρκ επίσης ε, αναφέρθηκε σε κάποιους κινδύνους οι οποίοι ψέρχονται. Απάντησα στα θέματα αυτά. Είναι θέματα εθνικής αρμοδιότητας κατά το διεθνέ δίκαιο. Ο κύριος Λόπος Αγγιλάρ. Συμφωνώ. Συμφωνώ με αυτά που είπατε ότι χρειάζεται ε, ένα σαφές, ένα σαφής δρόμος που θα μας οδηγήσει και πάλι στο Σέγγεν. Είχα ήδη πολλά προβλήματα με το Σέγγεν. Δεν θέλω να επανέλθουμε στα ίδια. Θα ήθελα να κρυθούμε προς τα εμπρός, να προχωρήσει ο χώρος Σέγγεν. Να καλωσορίσουμε τρία νέα κρατημέλη, αλλά και να λειτουργήσει καλύτερα ο χώρος Σέγγεν, η ζώνη Σέγγεν. Χρειάζεται λοιπόν ένας σαφής δρόμος Συμφωνώ απόλυτα. Είναι δύσκολα τα πράγματα βέβαια, να το πούμε και αυτό. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά στην τηλεδιάσκεψη την αυριανή με τους ε, Υπουργούς Εσωτερικών. Έχουμε αυτή λοιπόν την τηλεδιάσκεψη η οποία λάμβανε χώρα τρεις φορές την εβδομάδα, τώρα άπαξ εβδομαδιαίως. Αύριο λοιπόν θα συζητήσουμε τα θέματα της άρσης των συνοριακών περιορισμών και το πώς ε, θα επιτευχθεί η βαθμία. Πραγματικά ανυπομονώ να ακούσω και τις προτάσεις τους και τις ανησυχίες τους για τους εποχικούς εργαζόμενους. Ήταν σαφή οι κατευθυντήριες γραμμέ. εξ αρχής. Οι εποχικοί εργαζόμενοι θα πρέπει να επιτρέπεται να περάσουν τα σύνορα για να εργαστούν. Είναι σαφέ αυτό στι κατευθυντήριες γραμμέ. Ένα τελευταίο ερώτημα για το ηλεκτρονικό εμπόριο και για τι ηλεκτρονικέ υπογραφέ. Αυτό δεν είναι στον τομέα αρμοδιότητά μου πραγματικά. Δεν μπορώ να σας απαντήσω, λυπάμαι πολύ. Αλλά να σας διαβεβαιώσω ότι αναπτύσσουμε μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα αυτά και η κυβερνοασφάλεια και το εμπόριο αυτό θα είναι σημαντικό τμήμα του πακέτου. Σε αυτό μπορώ να επανέλθω ενδεχομένω, αλλά δεν είναι στο χαρτοπλάκι μου. Είναι ένα θέμα για τον Επιτροπό Ευχαριστώ. Pues muchísimas gracias. Eh, vamos ευχαριστούμε πολύ, λέει η Πρόεδρο. Και τώρα προχωρούμε δεύτερο γύρο ερωτήσεων από τους βουλευτές. Ποιος Κρίς Πίτερς είναι ο πρώτος. Ευχαριστώ. Ήδη έχετε απαντήσει πολλές ερωτήσεις και ελπίζουμε θα έχουμε και τις απαντήσεις σε αυτές όλες τις ερωτήσεις. Γιατί έχουμε αυτή την πρόσφατη ελληνοτουρκική κρίση στα σύνορα και αυτό ε, έχει σχέση με τις απάνθρωπες συνθήκες στους καταβλισμούς στα νησιά και έχουμε επαναλαμβανόμενα κάποιες ε, τραγωδίες και επίσης χρειάζεται κάτι να γίνει για άσυλο και μετανάστευση. Δεν είναι δυνατό να συνεχίσουμε να αναβάλουμε και έχω να σας ερωτήσω τα εξής τέσσερα. Πρώτε, πότε πρόκειται να υποβάλλετε κάποιες προτάσεις. Δεύτερον, τι μηχανισμοί αλληλεγγύης ε, σκέφτεστε ότι μπορεί να υπάρξουν μεταξύ κρατών μιλών γιατί με την κατάσταση ε, μεταναστών, ε, προσφύγων, των Επίσης, οι <clears throat> προτάσεις σας θα έχουν κάποιες διατάξεις συγκεκριμένες για τους ανηλίκους και επίσης για τον έλεγχο εσωτερικών συνόρων. Αυτοί οι περιορισμοί κατά τη γνώμη σας για τον κώδικα Σέγγεν ε, και επίσης ε, την οδηγία ελεύθερης διακίνησης ε, τι, τι, τι, τι, βλέπετε να γίνεται. Κυρία Σιλβί Γκυγιόμ, σας ακούμε, σας ακούμε. Γκυγιόμ, σας ευχαριστώ. καλημέρα σε όλους. Και εγώ θέλω να επανέλθω στο θέμα Σέγγεν. Το θέμα και η αρχή τη ελεύθερη διακίνησης είναι αδιαπραγμάτευτο. Θα πρέπει βέβαια να είναι τελευταία λύση με αντικειμενικά κριτήρια η έλεγχη. Τώρα περνάμε μια κρίση, οπότε έχουμε κατευθυντήρια της Ευρωπαϊκής επιπλέον για ελέγχους, για προσωρινή αναστολή, μη σκοπίμων μετακινήσεων. Ε, υπάρχει κάποια αναλογία και όλοι θα συμφωνείτε ότι τα κράτη-μέλη, το καθένα κάνει ό,τι ήθελε. Ε, υπάρχει μια αταξία από το 2015. Έχει γίνει η κατάσταση πολύ μπερδεμένη στο χώρο Σέγγεν. Έχουμε κινδύνους ε, για την ασφάλεια, πάρα πολλά κράτη-μέλη. Ε, επίσης ε, μονιμοποιούν τους ε, ελέγχους. Υπάρχει κατάτμιση στην Ένωση. Ε, αυτό δημιουργεί δυσπιστία από τους Ευρωπαίους προς την Ένωση. 55% ε, Γάλλων λένε ότι θέλουν και μετά την κρίση να κλείσουν τα σύνορα. Επίσης, ε, πιο απλό από πολιτική πλευρά είναι να υπάρχουν έλεγχοι παρά να αρθούν οι έλεγχοι. Κύριε Επίτροπε, τι θα γίνει. Θεωρείτε ότι η ενημέρωση μεταξύ κρατών μελών και με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το Σέγγεν ίσχυσαν και εσείς. Πώς θα συντονίσετε την άρση των μέτρων. Δεν πρέπει να υπάρχουν ε, μονομερείς ενέργειες ή θημερείς. Πότε να περιμένουμε να γίνει μια διοργανική συνεννόηση για το Σέγγεν. Νομίζω μέσω πρόθεσμα είναι σημαντικά όλα αυτά για να ξανακερδίσουμε την ε, εμπιστοσύνη των κρατών προς την Ένωση αλλά και του κόσμου. Κύριε Πτωδράτσε, ευχαριστώ. Και εγώ θα ρωτήσω κάτι για το Σέγγελο, κύριο Τουντοράτσε. Τα είπαμε και στην ομάδα μας. Να μην επαναλάβω όσα ελέγχθησαν. Τα περισσότερα που θέλω να σας πω, τα είπαν οι συνάδελφοι. Αλλά τα είπατε και εσείς στην αρχή Είπατε για συντονισμό, αποφυγή διακρίσεων, ε, τη της νομοθεσίας για το Σέγγεν και είπατε ότι θα υπάρξει την επόμενη εβδομάδα, αν κατάλαβα καλά, ανακοίνωση από πλευρά σας. Νομίζω θα πρέπει να διακρίνουμε ως κόκκινη γραμμή. Τι γίνεται, ποιος είναι ο ρόλος της Κομισιόν, τι γίνεται με το νομικό πλαίσιο. Τι διέπει το Σέγγεν. Θέλει η Κομισιόν, μπορεί από πολιτικής πλευράς να έρθει σε επαφή με τα κρατημέλη. Καλό είναι το ότι συνεχώς συνοείστε. Αλλά να μπορεί να είναι πιο αποφασιστική, πιο δυναμική για το Σέγγεν η Επιτροπή ως προς τα κρατημέλη. Το περιμένουμε αυτό τα τελευταία χρόνια. Θέλουμε να μας υποσχεθείτε ότι με ενεργό, με δυναμικό τρόπο θα κατοχυρώσετε το, το, το, το κεκτημένο. τι γίνεται τώρα. Συζητήσαμε και το πρωί για το Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε και απάντηση από το Ηνωμένο Βασίλειο και είμαστε μπερδεμένοι. Και εγώ και πολλοί άλλοι. Εσείς θα κάνετε κάτι, κάτι συγκεκριμένο τώρα. Τι μας λένε οι Άγγλοι ότι θα αγνοήσουν τις συστάσεις σας. Θέλουν τέσσερα χρόνια να εφαρμόσουν κάποιες άλλες συστάσεις. Μα τι θα γίνει. Μα έχουμε τέσσερα χρόνια από τότε που έγινε το δημοψήφισμα. Τώρα δεν υποχωρούν σε τίποτα. Θέλουν σχημένη συνεργασία, θέλουν δεδομένα, πρόσβαση αυτά, αλλά ε, θα πρέπει στη σχέση μας με τον Ρώμα Βασίλειο επιτέλους να είμαστε πιο αποφασιστικοί και θα πρέπει να δείξει πυγμή σε αυτό το μέτωπο η Κομισιόν. Τα είπατε για την εγκληματικότητα και ίδια, για την ε, ψηφιακή ταυτοποίηση, αλλά άρα χρειάζονται οι διοικητικές αρχές κάποια βοήθεια, χρειάζονται κάποιον στο πιδάλιο, δηλαδή Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα όλο ένα και περισσότερο έγκλημα θα έχουμε. Άρα Προσέξτε την εντολή της Europol. Περιμένουμε να αναβαθμιστεί η Europol φέτος. Να είστε φιλόδοξοι και σε αυτό. Και πρόεδρος. Κύριε Ερικ Μαρκάρ, μας ακούτε? Υπάρχει σύνδεση. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ε, πολλές ερωτήσεις που απαντήσατε ήδη. Έχω μια ερώτηση να κάνω. Λέτε πραγματικά ότι το θέμα στη Μάλτα και στη Μεσόγειο είναι θέμα τριτών χωρών οι άλλοι, δηλαδή έχουν μόνο την ευθύνη. Και τηλεφώνησα στις αρχές ε, στο σύστημα Μάλτα και ήταν πραγματικά δύσκολο να έχουμε επαφή. Το θέμα λοιπόν δεν ήταν να περιμένουν τρεις ημέρες. Και ενδεχομένως... Να πρέπει να σκεφτούμε και τι γίνεται και με τις ιδιωτικές, με τα ιδιωτικά σκάφη. Δεν ήταν θέμα δηλαδή μόνο ε, των αρχών της Μάλτας και θα χρειαστούν διευκρινήσεις εδώ. Υπήρχαν ε, κλιματικές ε, περιπτώσεις. Είναι δυνατόν όλοι τελικά δηλαδή να θεωρούν ότι δεν είναι υπεύθυνοι και να κατηγορούν τους άλλους. Μα ακούτε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριος Μουσάντε. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Έχω δύο ερωτήματα. Πρώτα-πρώτα, για το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου. Από ό,τι φαίνεται, εσείς υποχωρείτε σε κάποιους ε, βουλευτές που θέλουν να διευκολύνετε τους μετανάστες. Μα χωρίς να υπάρχει διάκριση, χορηγούνται κάποια επιδόματα σε όποιον έχουν ανάγκη. Μα τι γίνεται, γιατί έχουμε τώρα να καλύπτονται και οι παράνομοι και οι νομίμως διαμένοντες στην Ένωση. Οπότε, το αποτέλεσμα είναι το να δυναμητίζονται τα συστήματα υγείας. Έχουμε όλη αυτή την προσπάθεια δουλεμπορίου συμφωνούμε το ότι κοστίζει σε ανθρώπινες ζωές στην Μεσόγειο. Ε, κάντε πιο αυστηρό το νόμο. Πρόληψη, κυρώσεις για τους λαθροδιακινητές και επίσης για κάποιους ιδιωτικούς φορείς που συνεργάζονται. Δεν τους νοιάζει αυτούς τους ανθρώπους το ότι έτσι διαδίδεται η αρρώστια. Αλλάξτε ερώτα, συνειδητοποιήστε ότι η πολιτική μετεγκατάσταση έχει αποτύχει αυτό που χρειάζεται είναι αποτελεσματική έλεγχη. Χρειάζεται να ξέρουμε το πώς αυτοί οι άνθρωποι θα γυρίσουν στις χώρες τους. Να μπορέσουμε να κάνουμε και υγειονομικούς ελέγχους αυτούς που έρχονται. Και κάτι άλλο διαφορετικό. Ενημερώστε μας για τον κανονισμό Eurodac. Είμαι εισηγητής, ξέρετε. Όσον αφορά τα σχετικά δεδομένα, αυτό θα βοηθήσει και την αντιμετώπιση της ε, λαθρομετανάστευσης και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Τι γίνεται, νομίζω ότι έχει παγώσει τώρα η πορεία του νομοθετήματος. Ευχαριστούμε κύριε Αρβανίτη. Μας ακούτε. Υπάρχει σύνδεση καλή με τον κύριο Αρβανίτη. Κύριε Κώστα Αρβανίτη. Δεν μας ακούει. Ναι, μισό λεπτάκι. Κύριε Αρβανίτη, πατήστε το κουμπί. Okay. Thank you very much. Welcome. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι πάρα πολύ για την ενημέρωση και θέλω να μεταφέρω κιόλα και να ευχηθώ να ανταμώσουμε γρήγορα όλοι οι συνάδελφοι ξανά στο Ευρωκοινοβούλιο. Θέλω να πιστεύω ότι έχετε τι καλύτερε προθέσει για να βοηθήσετε την αντιμετώπιση τη κρίση. Όμω, αυτό που ζούμε σήμερα και στη δική μου χώρα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια διπλή πολιτική. Και θέλω να καταλάβω αν είναι διαφανή και ορατή η πολιτική στο προσφυγικό ή μήπω έχουμε μια παράλληλη υπόγεια πολιτική που εν τέλει κυριαρχεί. Τι εννοώ. Χθε έγινε η πρώτη συζήτηση στην Ελληνική Βουλή για το νομοσχέδιο στο προσφυγικό. Αυτό το νομοσχέδιο βοηθάει και επισπεύδει τη διαδικασία απόρριψη του ασύλου επιτρέπει τη δημιουργία κλειστών κέντρων κράτηση που δημόσια αποκηρύξατε. Θεσμοθετεί την κράτηση ακόμα και ανηλίκων. Χορηγεί μυστικά κονδύλια στο Υπουργείο για χρήση εντό και εκτό Ελλάδα χωρί καμία διαφάνεια. Θέλω επ' αυτού των μυστικών κονδυλίων, κυρία Γιώχαρσο, να μου απαντήσετε ακριβώ, αν το γνωρίζετε και ποια είναι η θέση σα. Θέλω να σα πω ακόμα ότι είπατε ότι υπάρχουν αλλαγέ στη λειτουργία του νομοσχεδίου στο Υπουργείο Μεταναστευτική Πολιτική και ότι είναι πραγματικό. Θα θέλαμε να μα πείτε αν είναι μια διαπίστωση και τι ακριβώ θέλετε να αλλάξει. Η κατάσταση στα camps αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι άθλια. Εν μέσω πανδημία έχουμε ουρέ για φαγητό και νερό, ανεπαρκή ενημέρωση των ετούντων για άσυλο για την κατάσταση, ανεπαρκή ιατρική φροντίδα. Θέλω να σα πω ότι το κονδύλι των 25 εκατομμυρίων ευρώ και η πρόβλεψη για 2.000 πρόσφυγε δεν έχει προχωρήσει ουσιαστικά. Μιλάω για το πρόγραμμα για τη φιλοξενία σε τουριστικά καταλήματα, που προχωράει με πολύ αργού ρυθμού, σαν να μην θέλει η κυβέρνηση να το προχωρήσει. Τι προτίθεστε να κάνετε γι' αυτό. Έχετε υπόψη σα ότι ο πραγματικό αριθμό των ανθρώπων μέσα και έξω από τι δομέ, μόνο στη Μόρια και τη Σάμμο, είναι τουλάχιστον δεκαπλάσιο. Και θέλω να σημειώσω και κάτι ακόμα. Τι θα κάνει ε, η Ευρώπη με τις χώρες που αρνούνται επισηματικά να παίρνουν μέρος στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης. Θα ζητήσετε κυρώσει, θα τις αφήσετε να χαράξουν δική τους πολιτική. Έγινε ένα πολύ μικρό βήμα θετικό, το στηρίξαμε, για τη μετεγκατάσταση των ανηλίκων. Πολύ ανεπαρκές και πολύ καθυστερημένα. Ακόμα και αυτή η πρωτοβουλία είναι γεμάτη ασάφεια. Σήμερα υπάρχουν στην Ελλάδα 5.500 ασυνόδευτα και εμείς μιλάμε για 50. Και εδώ έχουμε, δεν έχουμε πραγματική εικόνα είναι 50, είναι 51, είναι 48, είναι παιδιά που θα επανενωθούν με τις οικογένειες ή είναι αυτό που λέμε ασυνόδευτα παιδιά. Θέλω να επιμείνω στο θέμα αυτό της επιλογής των παιδιών. Είναι απάνθρωπο και προσβάλλει τις αξίες. Ποιος επιλέγει τα παιδιά. Φέρνει στο μυαλό μας ζωφαρές εικόνες σκλαβοπάζαρου. Και επιμένω πάλι και θέλω να κλείσω με αυτό, κυρία Γιώχανσον. Υπάρχει διγλωσία αυτή τη στιγμή. Και υπάρχει έλλειψη διαφάνειας. Επιμένω για το θέμα των μυστικών κονδυλίων και θέλω σαφή απάντηση επί του συγκεκριμένου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Κυρία Φεράρα, παρακαλώ, είσαστε συνδεδεμένοι. Πολύ καλά, μάλιστα. Το καλύτερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ε, Πίτροπε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Και θα ήθελα καταρχάς να μου δώσετε κάποιες διευκρινήσεις σε ό,τι αφορά το πακέτο ασύλου. Και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι τώρα είμαστε σε κατάσταση ανάγκης και έτσι δεν μπορεί εδώ να καθυστερούμε. Οπότε νομίζω ότι επίγει να ξεκαθαριστεί ποιες είναι οι προθέσεις της ε, Κομισιόν. Θα πρέπει να διατυπώσετε κάποιες προτάσεις, να δούμε τι νέα στοιχεία θα υπάρξουν και να ολοκληρωθεί αυτό, αυτή η προσπάθεια και από εμά και να πάει στο Συμβούλιο. Επίσης χρειάζεται υπό αυτήν την κατάσταση να δούμε το ότι ακόμα πολλές χώρες έχουν πρόβλημα όσον αφορά τη διαχείριση του προσφυγικού. Ιταλία, Μάλτα, Ελλάδα. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τώρα και τα δύο προβλήματα. Και την επιδημία και τις μεταναστευτικές ροές. Υπάρχουν ε, υγειονομικά πρωτόκολλα ευρωπαϊκά που να ενεργοποιηθούν τώρα σε σχέση με αυτές τις χώρες για τις μεταναστευτικές ροές. Επίσης, τι πρόγραμμα προτείνει υποτίθεται να προωθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτως ώστε να υπάρξουν εγγυήσεις για τις αρχές που κατοχυρώνονται στη συνθήκη για την κατανομή των ευθυνών. Είδατε τι έγινε στη Σάμο. Είχαμε αυτές τις ε, πυρκαγιές και ε, τώρα υπάρχει και το πρόβλημα της πανδημίας. Έχουμε το πρόγραμμα της μετεγκατάστασης των ενηλίκων, αλλά υπάρχουν και άλλοι που είναι ευάλωτοι και αυτοί θα πρέπει να καλυφθούν με κάποιες προτάσεις, κάποιες διατάξεις για να κατοχυρωθούν τα δικαιώματά τους. Τώρα για τη Λιβύη έχει γίνει πεδίο δοκιμής νέων όπλων. Παραδιάζεται το εμπάργκο του ΟΗΕ σχετικά με τη Λιβύη και προσπαθώ να καταλάβω ποιος είναι ο ρόλος της Ευρώπης. Τέρε τελειώνω. Ποιος είναι ο ρόλος της Ένωσης λέγω όσον αφορά την ε, βοήθειά της να υπάρξει ανακοχή και διάλογος ε, με τις ε, χώρες που μπορούν να μεσολαβήσουν μεταξύ των αντιμαχωμένο. Κυρία Γιώχανσον, αν μπορείτε απαντήστε για αυτό το δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Έχουμε κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις και κατόπιν να πάμε σε έναν τρίτο κύκλο, γιατί έχουμε τόσες ερωτήσεις προς εσάς. Μας ακούτε κυρία Γιώχανσον. Και έχετε το λόγο. Ναι, να προσπαθήσω να σας απαντήσω. Κύριε Πίτερς, όταν το συνεπότερο δυνατόν ολοκληρώσουμε το, το, το, το, νέο πλαίσιο, θα σας το παρουσιάσουμε. Άλλαξε τώρα το χρονοδιάγραμμα. Τα συζητάμε αυτές τις μέρες στην Κομισιόν. Και όπως ξέρετε, χρειάζονται συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε για να βγούμε από αυτήν την κρίση της πανδημίας. Λοιπόν, θα παρουσιάσουμε τις προτάσεις μας αρκετά σύντομα. Όταν γίνει αυτό θα τα πούμε. Ναι, θα καλύψουμε συγκεκριμένα τους ε, ανηλίκους. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα στα πλαίσια του μεταναστευτικού, το θέμα των ανηλίκων. λαμβάνεται υπόψη για όλα τα επιμέρους ζητήματα. Τι γίνεται για τους περιορισμούς τους, αν υπάρχει αναλογικότητα. Πολλοί, πολλοί βουλευτές ρώτησαν το ίδιο. Στην αρχή δεν υπήρχε αναλογικότητα. Είχαμε πολλά μέτρα ασυντόνιστα. Υπήρχε ένα κάποιο χάος όταν πρωτοκλείσαν τα σύνορα, αλλά σύντομα τα κράτη-μέλη κατάλαβαν ότι χρειάζεται περισσότερο συντονισμός, το ζήτησαν από την Κομισιόν, ζήτησαν κατευθυντήριε ε, και τώρα, όπως είπα στην αρχή, η κατάσταση κρίνεται σταθεροποιημένη. Θα ήθελα να είναι ακόμα καλύτερη, αλλά νομίζω ότι αρκετά καλά τα πάμε με την διαχείριση. Αυτό που κάναν τα κράτη-μέλη για τα σύνορα αντιστοιχεί κάπως αυτό που κάναν πάρα πολλοί άνθρωποι που σπεύσαν στα σούπερ μάρκετ, συσσόρευσαν χαρτιά τουαλέτας, κλείδωσαν τις πόρτες. Αλλά πάρα πολύ σύντομα κατάλαβαν ότι αυτό δεν λύνει το πρόβλημα. χρειάζεται συνεργασία και καλή γειτονία για αυτή την κρίση. Έτσι θα λυθούν προβλήματα και αυτό διαπιστώνουμε να υπάρχει τώρα. Άρα υπάρχει συνεργασία και αποδίδει. Ε, επίσης είπατε για διοργανικό θεσμικό διάλογο για το Σέγγεν. Αυτό είναι μια καλή πρόταση. Το πρότεινε κάποια βουλευτής. Ναι, ναι, θα το σκεφτώ σοβαρά. Κύριε Τουντοράτσο, ρώτησατε για το Ηνωμένο Βασίλειο. Μόλις από λίγες μέρες ολοκληρώσαμε μια σχετική έκθεση, ε, το Ηνωμένο Βασίλειο και όντως ε, ήταν πολύ ελλειπής ανεπαρκής. Η απαστερή θα πρέπει να αποκατασταθεί η κατάσταση γιατί χρειάζεται να δούμε το ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ποια θα είναι η μελλοντική μας σχέση. Και για τα θέματα ασφαλείας. Μα είπατε επίση ότι οι διοικητικέ αρχέ χρειάζονται καθένε γραμμέ, χρειάζονται επίση ενίσχυση, αναβάθμιση και επίση η εντολή προ την Europol. Ε, και αυτό το μελετάμε, να έχει πιο ισχυρή εντολή. Να δούμε πώς μπορεί να συνεργαστεί η Europol με ιδιωτικούς φορείς. Εταιρείες. Έχουμε τώρα στην Αμερική ένα hub, ένα κόμβο και υπάρχουν εκατομμύρια πληροφοριών σε σχέση με ιντερνετική κακοποίηση από πλευράς ε, εταιριών και στέλνουν τις πληροφορίες αυτές στην Europol από τις Ηνωμένες Πολιτείες και πάνε μετά στα κρατημέλη. Άρα, θα πρέπει σε αυτό το τομέα να δούμε πώς θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί στη δουλειά μας. Κύριε Μάρκερτ. Ναι. Θα σας καλύπτει και εσάς η καινούργια δεσμή με τον κύριο Μποξάντε. Ναι, θα πρέπει να καταπολύσουμε τις του τους λαθροδιακινητές. η διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν γιατί θα ενταθούν στη συνέχεια και μετά την κρίση. Υπάρχει όμως μία αντίφαση. Από τη μία θέλουμε να αποδεχτούμε μετανάστες και από την άλλη μεριά θέλουμε να βοηθήσουμε για την κρίση. Όμως, τι παρατηρείτε τώρα στις μέρες μας ότι θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την ε, επιδημία ε, τους ε, δουλε... αυτούς που δουλεύουν τέλο πάντων στα νοσοκομεία γιατί είναι πάρα πολλοί οι μετανάστες που δουλεύουν εκεί στον τομέα της υγείας άρα θα πρέπει να βοηθήσουμε και αυτούς Eurodac το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει βοηθήσει. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε γι' αυτό. Δεν θα αρχίσουμε από το Α, θα βασιστούμε σε αυτά που ήδη έχουν γίνει. Θέλουμε όμως κάποιες μικρές αλλαγές. Ας πούμε την πρωτοκόλληση, αρχιοθέτηση των αιτήσεων ε, και όχι μόνο των ετούντων, γιατί πολλές φορές ε, μία αίτηση καλύπτει ολόκληρη την οικογένεια και πολλές φορές ένα άτομο κάνει περισσότερες από μία αιτήσει. Άρα για τα στατιστικά χρειάζεται μία καλύτερη καταχώρηση. Κύριε Κωνσταντίνο Αρβανίδη, τι θα αλλάξουμε σε σχέση με αυτή τη δέσμη μέτρων. Θα σας τα παρουσιάσω, είπαμε βέβαια. Και ήδη απήντησα γιατί με την κατάσταση των πιο ευάλωτων από τα νησιά. Οφείλω να σας πω ότι δεν συμφωνώ ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι ε, ήδη είναι λίγοι αυτοί που έχουν μετεγκατασταθεί, ε, ότι είναι στα γονατό ωκεανό, μα για έφηβους και για παιδιά μικρά είναι πολύ δύσκολη η κατάστασή τους. Ε, υπάρχει φόβος για το μέλλον. Είναι πολύ σημαντικό το ότι μερικοί αυτού έχουν πάει σε κάποια κράτη-μέλη και κάνανε κάποια βήματα για το μέλλον του. Για μένα αυτό το οποίο έχει γίνει δεν είναι σταγόνα το κένο και είμαι πολύ περήφανη που κατάφερε η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει ε, πράξη την αρχή της αλληλεγγύης παρά το ότι τώρα είμαστε πάρα πολύ στριμωγμένοι από αυτή την ε, κρίση, αυτά τα επιπλέον προβλήματα που δημιούργησε ο ιός. Κύριε Φερέρα, όχι, όχι, κυρία Φερέρα, μας ε, είπατε για τις προτάσεις για την πανδημία. Ήδη εμείς έχουμε κάνει τις προτάσεις αυτές που λέτε τον Απρίλιο και τι να πω. Ναι, δεν έχουμε πει τίποτα για τη μετανάστευση αυτές τις προτάσεις, αλλά Συμφωνώ. Θα πρέπει να γίνει η κατανομή των ευθυνών. Είδαμε τι γίνεται σε Καναρία, Ιταλία, Μάλτα. Θα πρέπει κάτι να γίνει. Σε αυτά τα κρατημέλη που υφίστανται τεράστια πίεση μαζί με την πανδημία. Η γενική μας διεύθυνση προσπαθεί πάρα πολύ σκληρά. Να δούμε πώς θα έχουμε με την κατάσταση. Τι θα κάνουμε με κάθε αποβίβαση μεταναστών. Πώς θα μετεγκαταστήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Προσπαθούμε. Κάνουμε το καλύτερο. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε, λέει Πρόεδρος. Έχω να σας πω ότι στις ε, 4 και 14 λεπτά θα σταματήσουν οι αγορεύσεις. Άρα θα δώσω σε τέσσερις το λόγο από ένα λεπτό και να μπορέσει να απαντήσει η Κομισιόν. Αν μιλήσετε πάνω από ένα λεπτό, κλέβετε χρόνο από ένα συνάδελφο. Ρέσλερ, είστε εδώ. Είναι εδώ ο κύριος Ρέσλερ. Όχι. Καλά. Τι πω. Η κυρία. Κυρία Ντυπών. Αγαπητέ, αγαπητή Επιτροπή, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για τι πληροφορίε που μα δώσατε σήμερα και για την επισκόπηση τη δουλειά που πρέπει να γίνει ακόμα για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού. Μία ερώτηση να κάνω για πιο πολλές πληροφορίες. Για την εντολή. Αναφέρατε πού θέλετε να υπάρξουν ε, βελτιώσεις για την τρέχουσα θετία και την εντολή. Έχουμε ακόμα το ίδιο χρονοδιάγραμμα όπως πριν από το χρονοϊό. Μπορούμε να περιμένουμε λοιπόν μια νέα νομοθετική πρόταση στο δεύτερο μιση του έτους ή θα καθυστερήσει η πρόταση αυτή. Υπάρχουν πιο πολλές ιδέες για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε αυτή την εντολή. Η κυρία Γιόντσεβα, είστε εδώ. Έχετε συνδεθεί. Ναι, με ακούτε, η κυρία Γιόντσεβα. Ναι, σας ακούμε. Καταρχάς, να ευχαριστήσω. Μία ερώτηση έχω να κάνω για τη μετανάστευση. Πώς πιστεύετε ότι θα βοηθηθεί η Μάλτα. Τι θα αλλάξει με τη νέα σας πρόταση για τη Μάλτα, την οποία και ελπίζουμε να τη δούμε σύντομα. Για την μετανάστευση, οι μεταναστευτικές ροές. Μιλάμε για την πολιτική επαναπροώθηση κατάσταση. Θα πρέπει να βρούμε όμως, μια ισορροπία στη μετανάστευση. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν μια σωστή ανάλυση η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι παρούσα σε διάφορα τμήματα της Λιβύης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, προκειμένου να καταπολεμήσουμε τη μετανάστευση. Τρίτη ερώτηση για το Σέγγεν. Πώς μπορούμε να αναμένουμε μια στρατηγική ανάλυση για την τρέχουσα κατάσταση του Σέγγεν και το τι μπορεί να γίνει για να προστατευτεί η ζώνη Σέγγεν από απονομερείς δράσεις. Ευχαριστώ. Για Ζαν Κριστόφ Έτσεν. Είστε... Έχετε συνδεθεί? Όχι. Ο κύριος Φραντς. Έχετε σύνδεση? Όχι. Ο κύριος Βέιβερς. ο κύριος Μπρέιερ. Ο κύριος Βάιμερς. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Επίτροπε. Τους τελευταίους 12 μήνες ακούμε το εξής. Δυστυχώ υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση του κυρίου Βάιμερ και ε, δεν ακούγεται. Υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα, λέει η πρόεδρο. Να ακούσουμε τον κύριο Φραντ. Έχετε σύνδεση, παρακαλώ. Όχι. Ο κύριος Ουρμπάν Κρέσπο. Έχετε σύνδεση. Ευχαριστώ, λέγει ο Ζουρμπαν Κρέσπο. Κύριε Γιώργη, δεν έχουμε χρόνο. Μας είπατε για τους καταβλημούς των ε, προσφύγων. Εμείς αυτά τα θεωρούμε ως κέντρα κράτησης και θεωρούμε ότι είναι κάτι σαν ορολογιακή βόμβα γιατί δεν είναι δυνατόν και να υπάρχουν οι ελάχιστες υγειονομικές εγγυήσεις και μιλούμε για χιλιάδες ανθρώπους που είναι αθώοι, δεν έχουν κάνει έγκλημα, είναι ε, φυλακισμένοι. Κόβεται σύνδεση. Κόπηκε η σύνδεση. του και κόπια λέει και η πρόεδρος. Για να προσπαθήσουμε τώρα. Κυρία Γερόκα, μας ακούτε. Υπάρχει σύνδεση με την κυρία Γερόκα. Το κουμπί το κουμπί. Ευχαριστώ πολύ. Βλέπω ότι γνέφεται φατικά δεν ακούει τον εαυτό μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Επιτροπέ, που συμμετείχατε σε αυτή τη συνεδρίαση. Μεταξύ των άλλων ερωτημάτων για το θέμα τη μετανάστευση, θα ήθελα να θέσω κι εγώ ένα. Θα ήθελα να θέσω και ένα άλλο θέμα για άλλο χαρτοφυλάκι, το θέμα του trafficking, το θέμα τη διακίνηση. Έχω κάνει κάποιε προτάσει για τι γυναίκε που είναι θύματα διακίνηση. για να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα επανέλθουν στις αρχικές φρικτές τους συνθήκες. Θα πρέπει να φροντίσουμε τις γυναίκες αυτές. Έχουμε πολλές τέτοιες γυναίκες οι οποίες είναι αναλφάβητες. Δεν μπορούν να γράψουν, δεν μπορούν να διαβάσουν. Αυτά προωθούν με πλαιτικό πρόγραμμα η Επιτροπή για τα δικαιώματα των γυναικών και η Επιτροπή των Νομικών Υποθέσεων. Ζητώ την υποστήριξή σας. Έχουμε τέσσερα λεπτά για να απαντήσει η Επίτροπος Γιώχανσον. Έχετε το λόγο, δεν σας ακούμε ωστόσο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ καλή ανταλλαγή αυτή απόψεων και καταρχάς να πω ότι το θέμα της διακίνησης έχει ως σκόπο να προστατεύσει γυναίκες και παιδιά από το να έχουμε πιο πολλά θύματα. Προς την κατεύθυνση αυτή θα κάνουμε προτάσεις για το πώς θα προστατεύσουμε το Σέγγεν τώρα. Αυτά τα είπα και εισαγωγικά. Απάντησα διάφορες τέτοιες ερωτήσεις. Είναι δύσκολο το θέμα αυτό, αλλά σίγουρα είναι στην κορυφή των προτεραιοτήτων μου. Το αντιμετωπίζω καθημερινά πλέον. Ε, η κυρία Τυπώ για τη νέα νομοθεσία για την εντολή της Europol. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τη Europol σε ό,τι αφορά τις τρίτες χώρες, σε ό,τι αφορά τα κράτη-μέλη, σε ό,τι αφορά και τις επιχειρήσεις. Αυτό είναι το πεδίο εφαρμογή όπου θα πρέπει να ενισχύσουμε την εντολή της Europol. Επίσης, να τους δώσουμε πιο καλό εξοπλισμό για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το έγκλημα τη διακίνηση τις νέες μορφές κυβερνοεγκλήματος. Έχουμε λοιπόν το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν έχει ακόμα παρουσιαστεί, αλλά θεωρώ ότι θα είναι δυνατόν να παρουσιαστεί η νέα πρόταση για την εντολή της Europol, το τέταρτο Σα του Σας ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ για τη δυνατότητα αυτή που μου δώσετε να ανταλλάξουμε απόψε. Είναι πάρα πολύ εντατική η ανταλλαγή απόψεων και πολύ έντονη πάντα. Αλλά είναι πολύ ενθαρρυντικό το ότι ακούω και τη δεσμευσή σα και τι ε, γνώσει σα για το θέμα αυτό και την συμμετοχή σα στη δεσμευσή σα. Και προσβλέπω στην επόμενη ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψει. Ευχαριστώ. Muchísimas gracias, comisaria por Πάρα πολύ κύριε Επίτροπε για την ευαισθησία που δείχνετε και για τις προσπάθειες που καταβάλλετε και που έρχεστε τακτικά να μας τα πείτε. Ο Άμπας περισσεύει για ένα λεπτό. Και οπότε πρέπει να σας πω ότι η πρώτη τροπολογία την οποία ψηφίσαμε μαζί με την τροπολογία παρθμών ε, δύο γιατί πρόκειται για ταυτόσιμες απερίφθησαν. 31 ψήφι υπέρ και 36 κατά. Μηδέν ήταν οι εποχές. Ωραία. Ε, τότε να πάμε παρακάτω. Επόμενη ψηφοφορία. Η τελική ψηφοφορία του θέματος μας και τώρα θα πρέπει να διακόψουμε και να συνεχίσουμε σε άλλη αίθουσα, σε λίγα λεπτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους έλαβαν μέρος και πολλά συγγνώμη προς όποιους δεν μπόρεσαν να λάβουν το λόγο. Ελπίζω την να μην έχουμε τεχνικό πρόβλημα. Ευχαριστώ.